Καλό απόγευμα κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ήλθατε στη σημερινή συνεδρίαση. Κηρύττω την ε, έναρξή της. Έχουμε πολλές γλώσσες στη διάθεσή μας ως βουλευτές. Είναι βέβαια Δευτέρα απόγευμα. Γνωρίζετε ότι για πολλούς συναδέλφους είναι δύσκολο το να είναι εδώ Δευτέρα απόγευμα. Ελπίζω ότι θα έρθουν και άλλοι συνάδελφοι, όπως έγινε και στην προηγούμενη ακρόαση. Καλώς ήλθατε λοιπόν όλοι και θα ήθελα να κάνω δύο σύντομες παρατηρήσεις. Ανακοινώσει καταρχήν για το γλωσσικό καθεστώς έχω αναφερθεί ήδη και δεύτερον για τα έγγραφα είναι στη διάθεσή σας και επίσης η μαλλοντές στη διάθεσή σας και θα έχουμε μετάδοση στο διαδίκτυο. Έρχομαι τώρα σε σχέση με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να την εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη και περνάμε τώρα στα πρακτικά τα οποία σας έχουν διανεμηθεί. Εάν δεν υπάρξει κάποια αντίρρηση και αυτά μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί, Πάνω στο σημείο 3 ε, δημόσια ακρόαση για το ξέπλυμα χρημάτων και την φοροαποφυγή. Ποια θέματα γίνονται σε σχέση με τη συμμόρφωση και ποιοι είναι οι κανόνες και ποιοι τους εφαρμόζουν και πώς μπορούν να ελεγχθούν όλα αυτά. Αυτό θα είναι το πρώτο ήμιση της σημερινής συνεδρίασης, γιατί έχουμε διαιρέσει την ακρόαση σε δύο Καταρχήν θα ακούσουμε τις ευρωπαϊκές αρχές, εκπροσώπους των ευρωπαϊκών αρχών και γι' αυτό έχω το χαρά να καλωσορίσω τον κύριο Τζοβάνι Κέσλερ, ο οποίο είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΟΛΑΒ, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Δίωξης της Απάτης. Επίσης τον Σίμα Ορίοντε, ο οποίος είναι ε, εκπρόσωπος, εκπρόσωπο εκπρόσωπος Europol και του δικτύου FIU της Europol. καλώ ήρθατε. Καθώς και τον Κλάου Μέιερ Κάμπρι, ο οποίος είναι Γερμανός μέλος του σώματος Eurojust. Και πρωτού ξεκινήσουμε, θα ήθελα να κάνω τις ε, υπομνήσεις. Είναι η τέταρτη ακρόασή μας σήμερα <clears throat> και προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια συνολική εικόνα και να κάνουμε τις απαραίτητες προετοιμασίες ώστε να έχουμε ένα πρώτο έγγραφο εργασίας. Έχουμε συζητήσει για, τις, για τα διεθνή πρότυπα σε σχέση με τα θέματα αυτά. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργούν οι διάφοροι εποπτικοί φορείς οι οποίοι προβλέπονται από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη του ξεπλήματος χρημάτων και εναντίον των φορολογικού χαρακτήρα απατών. Θα θέλαμε λοιπόν καταρχήν να ελέγξουμε ποια είναι τα απαραίτητα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν και τι προκύπτει από την νομοθεσία, την τρίτη και τέταρτη οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος, πώς μπορούν να εφαρμοστούν καλύτερα αυτές οι νομοθετικές πρόνοιες σε σύνδεση και με τα προβλήματα που ανέδειξαν τα έγγραφα του Παναμά. Τρίτο σημαντικό σημείο επίσης θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις για το περαιτέρω έργο μας ως ε, συμπεράσματα από τις ακροάσεις που διεξάγουμε. Σας είπα ότι έχουμε δύο τμήματα της ακρόασης. Το πρώτο πάνελ θα ακούσουμε τις εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Φορέων, ενώ στο δεύτερο πάνελ θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά από μια εθνική οπτική γωνία. Έχουμε εκπροσώπους από τα εθνικά κράτη. Αλλά θα ήθελα επίσης να να σας πω ότι ότι έχουμε την μονάδα FATF, Financial Action Task Force, δηλαδή τη μονάδα για δράση στα χρηματοπιστωτικά. Είναι ένας φορέας ο οποίος βρίσκεται υπό την αιγίδα της Κομισιόν και που παρακολουθεί τις παγκόσμιες εξελίξεις στο ξέπλυμα χρημάτων και στα θέματα φοροαποφυγής. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε κάποιος ο οποίος να είναι έτοιμος να έρθει στην ακρόασή μας. Επομένως, την προηγούμενη εβδομάδα ήρθα σε επαφή με τον πρόεδρο αυτού του φορέα, ζητώντα σε μία από τις μεταγενέστερες ακροάσεις μας να υποδείξει κάποιο άτομο το οποίο μπορούμε να προσκαλέσουμε. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί και η Κομισιόν σε πολλές από τις ε, προτάσεις της χρησιμοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της FATF. Δεύτερον, έχουμε προσκαλέσει την, ε, ε, την επιθεώρηση για τα χρηματοπιστωτικά θέματα από την Σουηδία για να συμμετάσχει στις ακροάσεις μας, αλλά μας είπαν ότι η χρηματοπιστωτική αυτή υπηρεσία ελέγχου έχει αυτή τη στιγμή να παρουσιάσει το έργο της ενώπιον της ειδική Επιτροπής που θεσπίστηκε στο Σουηδικό Κοινοβούλιο, κάτι το οποίο αποτελεί νομική υποχρέωση αυτή και μόνο μετά θα μπορέσει να έλθει ενώπιον μας και είπανε ότι δεν μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες ή πιο πριν να δώσουν πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ό,τι στο Σουηδικό Κοινοβούλιο. Τρίτον, οι Σουηδικές ε, αρχές που είναι αρμόδιες για τα θέματα αυτά, οι οποίες είχαν ε, παρουσιάσει πληροφορίες που αφορούν περίπου 560 δανούς φορολογούμενους για ποσά φοροαποφυγής που φτάνουν περίπου τα 6 εκατομμύρια δανεικές κορώνες, 800.000 ευρώ, είναι τώρα στη φάση της διενέργειας ερευνών σε σχέση με τα άτομα αυτά και τις ε, εταιρείε και μας είπαν ότι όταν προχωρήσει αυτή η διαδικασία μόνο τότε θα είναι σε θέση να έρθουν ενώπιόν μας. Αυτά λοιπόν και έτσι βλέπετε ότι πέραν των σημερινών καλεσμένων Εμεί προσπαθήσαμε να έχουμε και περαιτέρω ε, καλεσμένους οι οποίοι θα έρθουν ενώπιόν μας στι επόμενες ε, συνεδριάσεις μα. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθω στου τρει ομιλητέ μα. οι οποίοι σα είναι και πολύ καλά γνωστοί, ο Τζοβάνι Κέστερ ο Γενικός Διευθυντής της Όλαφ από το 2011. Καταρχήν, ο κύριος Κέσσερ υπήρξε εισαγγελέα στην Ιταλία προτού γίνει ε, επικεφαλής τη ΟΛΑΦ. Είναι καταρχην ο κύριο εδώ γιατί είχαμε πολλές συζητήσεις μαζί του και στο παρελθόν και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας κύριε Κέσλερ. Στη συνέχεια θα επανέλθω στον κύριο Ριοντέ από τη Γαλλία εκπρόσωπο της ε, Europol, καθώς και τον Κλάους Μάιερ Κάμπρι από την Eurojust από την Γερμανία. Μέλος του Eurojust από τη Γερμανία. Οι κανόνες μας είναι ως εξής, όπως συμφωνήσαμε. Υπήρξαν κάποια ερωτήματα τα οποία δόθηκαν γραπτά στους ομιλητές, τα οποία τα έχουν απαντήσει. Μας δόθηκαν τελευταία στιγμή απαντήσεις και αυτό διότι ήταν αργία η Παρασκευή στο Βέλιο. Θα έχει ο κάθε ομιλητής 10 λεπτά για, εισαγωγικές, για εισαγωγική ομιλία και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων σε χρονοθυρίδες 5 λεπτών με κάθε μέλος του πάνελ. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Κέστα. Έχετε το λόγο κύριε Κέστα. Uh, Αγαπητά μέλη, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας <clears throat> σε αυτήν τη δημόσια ακρόαση. Να αναφερθώ σε αυτά τα οποία κάνει, έχει ήδη κάνει η Όλαφ για τον φάκελο που έχετε μπροστά σας. και για τις προτάσεις της πολιτικής φύσεως που έχουν γίνει για τη συνέχιση των εργασιών μας. Εμείς ελέγχουμε απάτες και παρατυπίες που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Ασχολούμαστε επίσης και με παράνομες συμπεριφορές του προσωπικού των θεσμικών οργάνων. Έχουμε ανακριτικές διαδικασίες και έχουμε επίσης και ε, εντολή στην, να συνεισφέρουμε αν θέλετε στη διαμόρφωση της στρατηγικής καταπολέμησης της απάτης. Στα πλαίσια της διερευνητικής μας δραστηριότητας χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες ελεύθερης πηγής οι οποίες είναι διαθέσιμες. Έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα για να αναλύουμε και να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που προέρχονται από τα λεγόμενα open source. Όταν δημοσιεύθηκαν τα Panama Papers λοιπόν, εμείς ε, αναλύσαμε κάποια στοιχεία και είπαμε ότι θα είχε και ενδιαφέροντα τμήματα για την καταπολέμηση ε, της ε, διαφθοράς και την καταπολέμηση παράτυπων συμπεριφορών του προσωπικού της Ένωσης. Αυτή στιγμή λοιπόν τα έγγραφα έγιναν διαθέσιμα. Εμείς ε, τα συγκεντρώσαμε όλα αυτά τα στοιχεία, τα κατεβάσαμε 430.000 ε, ε, θα έλεγα καταχωρήσεις ή ονόματα καταχωρήσεων, προσώπων, εταιριών, επιχειρήσεων, ό,τι ήταν διαθέσιμο. Ε, εμείς προσπαθήσαμε να δούμε αν οι, τρεις, οι εξής τρεις κατηγορίες συνδέονται με τις εταιρείες αυτές τις offshore οι οποίες περιλαμβάνονται στα Panama Papers. Τρεις είναι οι κατηγορίες που μας ενδιαφέρουν. Καταρχάς, προσωπικό και μέλη των θεσμικών οργάνων, θα σας το αναλύσω αυτό. Δεύτερη κατηγορία, εμπειρογνώμονες που παρέχουν υπηρεσίες στα πλαίσια κοινοτικών προγραμμάτων και άνθρωποι οι οποίοι ωφελούνται από τα κοινοτικά κονδύλια. Και τρίτον, πρόσωπα ή φυσικές οντότητες που έχουν ήδη έρθει σε γνώση της Όλαφ σε προηγούμενες έρευνες της. Λοιπόν, τρεις κατηγορίες, θα επανέλθω σε αυτές. Εμείς τι κάναμε. Ελέγξαμε αν στις 430.000 καταχωρήσεις, ονόματα, επιχειρήσεις κτλ. Υπάρχει μια κάποια σχέση με ανθρώπους που ανήκουν στις τρεις κατηγορίες τις οποίες προανέφερα. Κάναμε την απαραίτητη έρευνα λοιπόν, ελέγξαμε αν στις 430.000 που ήταν διαθέσιμες υπήρξαν μέλη του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, τι είδους προσωπικό ήταν αυτό. Εμείς συγκρίναμε τα στοιχεία και με το δικό μας σύστημα Ασχοληθήκαμε επίσης με τα ονόματα όλων των επιτρόπων, όσων υπαλλήλων είχαν υψηλού επίπεδου διαχειριστικές θέσεις, ε, ονόματα γενικών διευθυντών, μεταξύ των οποίων και το δικό μου, ε, ονόματα των γενικών διευθυντών και των εκτελεστικών διευθυντών των περιφερειακών οργάνων, τα μέλη όλων, ε, τα μέλη τα κοινοβουλευτικά, τα ονόματα των κοινοβουλευτικών μελών, που αλλάζουν τα τελευταία χρόνια ε, και γενικά ό,τι είναι δημόσια διαθέσιμο. Και ταυτόχρονα συμπεριλάβαμε και τα ονόματα των κατηγοριών του προσωπικού που θεωρούνται ότι εκτίθενται σε υψηλούς κινδύνους. Προσωπικό για το οποίο υπάρχει ένα ξεχωριστό ε, πλαίσιο λειτουργίας και ανεξαρτησίας. Σαν παράδειγμα, δημοσιονομικοί υπόλογοι, διατάκτες, ελεγκτές, όλα τα ονόματα αυτά λοιπόν τα συγκεντρώσαμε και τα ελέγξαμε απέναντι στα ονόματα τα οποία είχαμε μέσω των 430.000 ξαναλέω καταχωρήσεων των Panama Papers. Η δεύτερη κατηγορία δεδομένων λοιπόν, όπως είπα, ήταν αυτοί που παρέχουν σαν εξωτερικοί συνεργάτες υπηρεσίες σε κοινοτικά προγράμματα και αυτοί που ωφελούνται και εισπράττουν κοινοτικά κονδύλια. Και τέλος, πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται ε, στις ε, παλαιές αλλά και τρέχουσες έρευνες της ΟΛΑΦ στόχος μας δεν ήταν να ανακαλύψουμε νέες απάτες εις βάρος των δημοσιονομικών της Ένωσης ή ε, απαράδεκτες συμπεριφορές μελών ε, των ευρωπαϊκών οργάνων, αλλά να προσπαθήσουμε να δούμε σε ποιες πλευρές η δράση μας και η λειτουργία μας παρουσιάζει ε, σημεία τροτά για να προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε καλύτερα στο μέλλον. Λοιπόν, εμείς ελέγξαμε 40.000 ονόματα προσώπων και επιχειρήσεων που ανήκουν στις τρεις κατηγορίες που προανέφερα. Το 60 περίπου 100 αυτών των 40.000 συνδέονται με την τρίτη κατηγορία, δηλαδή πρόσωπα και ε, εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται ήδη ε, σε έρευνες τις οποίες έχει κάνει ή συνεχίσει να κάνει η ΟΛΑΦ. Ελέγξαμε λοιπόν να δούμε αν οι 430.000 αυτές καταχωρήσεις των Panama Papers αφορούσαν και σε ανθρώπους ή επιχειρήσεις ή οντότητες ε, ανθρώπων ή εταιριών που έχουν σχέση λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ένα τρόπο ή τον άλλο. Η προσπάθεια που έγινε λοιπόν ε, δεν ήταν εύκολη. Υπήρξε καταρχάς ένας καθαρισμός των δεδομένων. Ε, μπορέσαμε δηλαδή εμείς να αντιμετωπίσουμε κάποιες ασυμβατότητες που υπήρχαν υπήρχαν προβλήματα μετάφρασης από το κυριλικό στο ε, λατινικό αλφάβητο και τέτοιου είδους δυσκολίες έπρεπε όλα να τα κάνουμε ξεκάθαρα και συγκρίσιμα. Και τέλος αυτά τα 40.000 ονόματα τα ε, βάλαμε σε μια νέα βάση δεδομένων. Ε, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε ακριβώς τις καταχωρήσεις αυτές και είδαμε τι αυτόματες προσωμιώσεις υπήρχαν στις καταχωρήσεις των Panama Papers. Υπήρξε ε, λίγο μικρός αριθμός ανθρώπων που συνέπεσαν και στις δύο κατηγορίες. 40.000 από τη μία, 340.000 από τη μία και τελικά ταυτίζονται 17. Βλέπουμε πολύ μικρός ο αριθμός αυτός. Εμείς ελέγξαμε χιλιάδες κόσμο και φτάσαμε σε 17 μόνο και αυτό είναι ένα καλό μήνυμα για τα ευρωπαϊκά όργανα. πολλά από αυτά τα στοιχεία α, ήδη ελέγχονται από την ΟΛΑΦ πριν δημοσιευθούν τα Panama Papers. Το 50% περίπου των 17 αυτών συμπτώσεων ήδη είναι επιχειρήσεις ή πρόσωπα φυσικά που ήταν ή είναι ε, υπό έλεγχο από την ΟΛΑΦ. Και αυτά βέβαια ήταν ενδιαφέροντα για τις ε, υποδιαξαγωγή ερευνές μας. Επί τη βάση λοιπόν της αναλύσεως την οποία σας παρουσίασα και επί τη βάση συμπληρωματικών στοιχείων πληροφορίας που συνδέονται με τα Panama Papers, τα οποία όμως συνελέγησαν από άλλες ε, ε, πηγές, ξεκινήσαμε τέσσερις διαδικασίες έρευνας. Ε, είναι σε εξέλιξη και δεν μπορώ να σας δώσω καμία επιπλέον πληροφορία για αυτές. Να πω ότι όλα αυτά εξετάζει τα θέματα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι ε, ένοχα. Εμείς σεβόμεθα την προϋπόθεση αθότητας. Να πω επίσης ότι εμείς χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία τα οποία ήταν δημόσια διαθέσιμα ενώ στα Panama Papers υπάρχουν πολύ περισσότερα στοιχεία. Εμείς αυτό το οποίο μπορέσαμε να ελέγξουμε ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν άλλες περίπου 11 εκατομμύρια υποστηρικτικά κείμενα τεκμηρίωσης, τα οποία δεν είναι ακόμα διαθέσιμα. Δεν είναι διαθέσιμα ούτε σε μας και ούτε και σε κανέναν άλλο από ό,τι ξέρω περιλαμβάνονται εξουσιοδοτήσεις προς δικηγόρους, επίσης πάρα πολλά ηλεκτρονικά ταχυδρομεία που αναφέρονται στους τελικούς ιδιοκτήτες, χρήστες αν θέλετε, ε, που προσπόρησαν κέρδη από τις επαγγελματικέ αυτές τοποθετήσεις. Λοιπόν αυτά για την Όλαφ, το τι έχει κάνει η Όλαφ. Τώρα να αναφερθώ λίγο σε κάποιες σκέψεις περισσότερο πολιτικής φύσεως. Τα ευρωπαϊκά όργανα υιοθέτησαν το 2015 την οδηγία για την καταπολέμηση ε, της ε, παράνομης ε, οικονομικής δραστηριότητας, της, του προσπορισμού ε, ποσών από παράνομες δραστηριότητες και περιμένουμε μέχρι το τέλος του 2016 να μεταφερθεί η οδηγία αυτή στις εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτό το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Ήδη τον Ιούλιο του 2016 προτάθηκαν κάποιες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροπολογίες έτσι ώστε να αλλάξουν οι αρμοδιότητες και εξουσίες των ερευνητικών υπηρεσιών στον τομέα αυτό ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να ελέγχουν πλέον τις συγκεντρωτικές τράπεζες δεδομένων όπως επίσης και την κίνηση των κεντρικών λογαριασμών έτσι ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε ευκολότερα τους πραγματικούς και τελικούς ιδιοκτήτες και χρήστες των τραπεζικών λογαριασμών. Λοιπόν αυτό το οποίο θα ήθελα εδώ να προσθέσω είναι ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις βέβαια αλλά από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να πω ότι η εμβέλεια όλων αυτών είναι περιορισμένη. Είναι σημαντική ότι η έκπλυνση σε εισαγωγικά χρήματος ε, και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Το θέμα είναι όμως να ανοιχνεύσουμε τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες που στρέφονται σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε ένα επιπλέον βήμα. Αν πρέπει εμείς να δημιουργήσουμε ένα εθνικό μητρό εθνικών λογαριασμών θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένο, εύχριστο και όχι διαθέσιμο μόνο στις υπηρεσίες έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε όλες τις άλλες εμπλεκόμενες κατασταλτικές υπηρεσίες. Και κατά τη διάρκεια της έρευνας θα πρέπει να υπάρχουν έρευνες ε, για όλες τις οικονομικές παρανομίες. Γιατί μόνο για την φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή, την έκπληνση βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Είναι λίγο τεχνικός ο διαχωρισμός και υπάρχουν και άλλες ε, οικονομικές συμπεριφορές παράνομες. Πολλές φορές όλες αυτές οι κατηγορίες, οι εγκληματικές, οι ποινικά κολάσιμες είναι διασυνδεδεμένες. Και γι' αυτό λοιπόν είναι δύσκολο να τεκμηριώσει κανείς το γιατί του ισχύοντος διαχωρισμού σήμερα. Υπάρχει μια οδηγία για την τρομοκρατία, κάνουμε ότι μας λέει οδηγία. Υπάρχει μια οδηγία ε, για ε, τις ε, παράνομες οικονομικές δραστηριότητες και μεταξύ τους διαφέρουν και κάθε μία οδηγία αλλού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν κύριε Κέσλερ που μας ε, παρουσιάσατε το τι κάνει η Όλαφ. Μας δώσατε και αριθμητικά στοιχεία. Τα πράγματα δεν είναι τόσο εκτενή, αλλά θα συνεχίσουμε να σας ε, θέτουμε ερωτήματα. Καλύτερα έτσι, καλύτερα ποιότητα παραποσότητα. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Σιμών Ριοντέ από τη Πόλο. Άξιτε με Πρόεδρε, και αξιότιμοι βουλευτέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που καλέσατε τη Europol στι 3 Απριλίου 2016. Η Διεθνή Επιτροπή ε, Δημοσιογράφων Ερευνητών απεκάλυψε στοιχεία για την ε, ύπαρξη δεδομένων που είχαν διαρρεύσει από τι ιστορικέ υπηρεσίε, από του ιστορικού σερβέρ τη νομική υπηρεσία Mossack Fonseca. Και τα ε, πρόκειται για 11 περίπου 5 εκατομμύρια στοιχεία και φακέλους, περίπου 2,6 τεραμπάτ που καλύπταν χρονική περίοδο περίπου 40 χρονών, χρόνων από το 1977 μέχρι το 2015 και περιλαμβάνουν ε, χιλιάδες ε, νομικά και φυσικά πρόσωπα. Αυτό στην συνέχεια θα το αναφέρουμε ως τα ε, Panama Papers. Στις 9 Μαΐου 2016 το σώμα αυτό δημοσίευσε στο κοινό μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει περίπου 3.200.000 εταιρείε, συγγνώμη, 320.000 εταιρείε οι οποίε αποτελούν τμήμα των Panama Papers και ονομάζονται Offshore Leaks. Και έχουμε λοιπόν και τη βάση δεδομένων για τα Panama Papers. Η ακριβή ε, διαδικασία δημιουργία τη βάση δεδομένων για τα Panama Papers δεν είναι σαφή και φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν κάποια εσωτερικά ε, αρχεία που ανήκαν στη Μόζακ Φοντσέκα και δεν αποτελούσαν αποτέλεσμα τη ανάλυση των συνολικών αυτών φακέλων. Με δειγματοληπτικού ελέγχου, στην βάση δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι κάποιες οντότητες που είχαν ε, συνδεθεί από τα μέσα με τα Panama Papers δεν ε, εμφανίζονταν στη βάση δεδομένων που αφορούσαν τα θέματα αυτά. Επίσης δεν υπάρχει πληροφορίες ε, για τις ε, λογαριασμούς τραπεζών, για την ε, επικοινωνία και για τις πληροφορίες τις σχετικές. Ωστόσο, η Europol κατέβασε την βάση δεδομένων Panama Papers και έκανε έλεγχο για να εντοπίσει τις κοινέ οντότητες και τα αποτελέσματα λοιπόν ήταν τα εξή. Έχουμε 3.469 τέτοιες ε, φακέλους και μάλλον τέτοιες κοινέ εταιρείε και ε, αποστάλησαν τέτοια πακέτα χωρών. Έχουμε λοιπόν 1722 ε, τέτοια στοιχεία τα οποία εντοπίστηκαν. Και έχουμε και το EOC στην ε, εντοπίσε 516 τέτοιες ε, περιπτώσεις και ενδεχομένως να υπάρχει λοιπόν μια σύνδεση με τους ρωσόφωνους και τις υπηρεσίες ε, της εταιρείας Μοσάκα Έχουμε επίσης ε, και το focal point Indra στην έκτη θέση σε ό,τι αφορά τον Ισλαμικό τρομοκρατία με 116 τέτοιες, ε, τέτοια ευρήματα. Και το βασικό είναι να γίνει σύνδεση των εταιριών από το Panama Papers, όχι μόνο με οικονομικά εγκλήματα όπως το ξέπλυμα χρήματος και διαφυγή ΦΠΑ, αλλά και με την τρομοκρατία, τη ρωσική τρομοκρατία, το κυβερνό έγκλημα και το καθεξής. Και πρέπει να πούμε ότι το Ηνωμένο Βασίλη ήταν η χώρα η οποία ε, είχε τα πιο πολλά hits, 1377, ε, αλλά αυτό θα μπορούσε να προκύπτει και από το γεγονό ότι αυτοί ήταν που έδωσαν τα πιο πολλά στοιχεία στο Focal Pay Point Sistrans. Η Λιθουανία ήταν στην τρίτη θέση γιατί είχε επίσης μεγάλη παρουσία ρωσοφωνών. Κάποιες ημέρες μετά λοιπόν τα Panama Papers και την δημοσίευση στα μέσα ενημέρωσης, η Europol ζήτησε από όλους τους εταίρους αν σκοπεύουν να ξεκινήσουν έρευνες σε σχέση με τα Panama Papers και Κάποιες χώρες απάντησαν θετικά και πολλές ε, έδειξαν διάθεση να ξεκινήσει έρευνα σε περίπτωση που υπήρχαν σχετικές ενδείξεις. Και επίσης ε, και η Europol συμμετείχε στη συνάντηση της Eurojust για τις ε, έρευνες στα κράτη-μέλη. Δυστυχώς, τα βάση δεδομένων Panama Papers και οδήγησαν σε πολλές χώρες σε έρευνες και άρνηση όμως του ICG να ξεκινήσει τέτοιες έρευνες. Η Europol δεν είναι σε θέση, δεν έχει ε, στην κατοχή της τα δεδομένα των Panama Papers. Μόλις τα έχουμε στη διάθεσή μας θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να ερευνήσουμε τις σχετικές ροές και να κοιτάξουμε με τα πολλά αυτά δεδομένα τι θα γίνει και θα συνδεθεί αυτό με πολλές ε, offshore εταιρείε. Είναι στη διάθεση των κρατών μελών λοιπόν η Europol για να συνδράμε στις σχετικές έρευνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ρέντε. Και τελευταία παρατήρηση ήταν πράγματι, πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί δεν έχουμε εμείς ακόμα πλήρη πρόσβαση. Θα εξαγάγετε φυσικά τα απορίσματά σας από τις έρευνες και είναι επικίνδυνο πολύ ενδιαφέρον ότι έχετε πάνω από 3.400 hit και τα σημεία εστίαση τα οποία αναφέρατε. Σας ευχαριστώ. Και τρίτος εμπειρογνώμονα είναι ο κύριος ε, Κλάου Κάπρι, που είναι Γερμανός από την Επιτροπή Eurojust. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Ίσως αυτά θα είναι τα τελευταία μου λόγια στα γερμανικά. Αλλά ως ε, αντιπρόεδρος της ε, Europol θα πρέπει να χρησιμοποιήσω την επίσημη γλώσσα αυτού του φορέα, δηλαδή την αλβιονική. Και γαλλικά θα μπορούσε, λέει ο κύριος Κάμπρη. Πρώτα απ' όλα, να κάνω μια εισαγωγή για τον λόγο της Eurojust στα θέματα ξεπλήματος χρήματος και μετά θα έρθω στα σημεία όπου έχουμε εντοπίσει νομικά προβλήματα αλλά και πρακτικά προβλήματα συνεργασίας. Η Eurojust, όπως ξέρετε, είναι η ομάδα δικαστικής συνεργασίας και ο στόχος μας είναι να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε το συντονισμό των ερευνών που γίνονται καθώς και των δικαστικών διώξεων και φυσικά να έχουμε την ε, συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων αρχών. Η συνεργασία μέσω του συντονισμού είναι το σύνθημά μας. Αυτό δεν αφορά μονάχα τα κράτη-μέλη, αφορά και τρίτους φορείς, στην περίπτωση αυτή τον Παναμά, που είναι ένας ε, εταίρος συνεργασίας σε αυτήν την περίπτωση. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε ότι εργαζόμαστε επί τη βάση αιτήσεων από τις εισαγγελικέ αρχές κρατών μελών. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μία ε, έρευνα με δική μας πρωτοβουλία. Ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε για την ε, <clears throat> εργασία αυτή. Καταρχήν έχουμε τις συναντήσεις συντονισμού. Οι συναντήσεις αυτού, αυτές σε απλά λόγια σημαίνει ότι φέρνουμε από κοινού όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, τις εθνικές εισαγγελίες ή τα δικαστήρια, τις αστυνομικές δυνάμεις και συζητούν μια περίπτωση από την αρχή ως το τέλος. Συμφωνούν για το πρακτέο, συμφωνούν για τα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν και φυσικά υπάρχει επιμερισμός των διαθεσίμων πληροφοριών. Το πιο σημαντικό για αυτέ τι συναντήσει είναι ότι δημιουργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνη μεταξύ των εισαγγελικών αρχών των διαφορών χωρών που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνεργασία του. Επίση έχουμε τα κέντρα συντονισμού, τα οποία είναι κέντρα στα οποία οργανώνονται κοινέ δραστηριότητε, μέρε δράση σε μια συγκεκριμένη μέρα, σε μια συγκεκριμένη περιοχή γίνονται <clears throat> κοινά μέτρα παραγωγός χάρη ε, έρευνες σε κατοικίες, συλλήψεις υπόπτων κτλ. Και επίσης υποστηρίζουμε τη διενέργεια κοινών ερευνών από κοινέ ομάδες έρευνας και ανάκρισης. Αυτές είναι ομάδες οι οποίες απορρέουν από συμφωνημένες ενέργειες και ανοίγουν το δρόμο για επιμερισμό πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Πώς εμπλέκεται τώρα η Eurojust στα θέματα ξεπλήματος χρήματος. Εμείς έχουμε δει να αυξάνεται σημαντικά από το 2012 ο αριθμό των περιπτώσεων. Είχαμε 148 περιπτώσεις το 2012 για ξέπλυμα χρήματος. Τώρα είμαστε στις 285 και συνεχίζεται ακόμα η χρονιά. Σύμφωνα εδώ απόλυτα με τον Τζοβάνι Κέσλερ, το ξέπλυμα χρημάτων είναι ένα οριζόντιο αδίκημα. Έχει να κάνει με την απάτη, με τη διαφθορά, με οργανωμένες ε, ομάδες εγκλήματος, με λαθρεμπορία ανθρώπων και με τρομοκρατία. Είναι κάπως λοιπόν <clears throat> τεχνητό να διαχωρίσουμε σε κατηγορίες όλα αυτά τα θέματα. Στις περιπτώσεις που έχουμε δει, σε 57 συναντήσεις συντονισμού, συζητήθηκαν θέματα ε, για το ξέπλυμα χρημάτων και δημιουργήθηκαν 12 ειδικέ ομάδες για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Σε 57 λοιπόν συναντήσεις συντονισμού για τις 285 περιπτώσεις. Αυτό σας δίνει την ε, γενική ιδέα για το πόσο σημαντικός είναι ο συντονισμό αυτός. Περίπου το 1 τέταρτο όλων αυτών των περιπτώσεων εμπλέκει μια διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση του. Ποια είναι τα προβλήματα λοιπόν που έχουμε αντιμετωπίσει και πώς θα μπορούσαν να επιληθούν τα προβλήματα αυτά. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις για την εκπλήρωση των αιτήσεων αμοιβαία αρρωγής. Πολλές φορές είναι χρονοβόρα αυτή η διαδικασία και απαιτεί και επιπλέον αιτήσει για τραπεζικούς λογαριασμούς, για κατοχή στοιχείων ενεργητικού, παραγωγός χάρη εγγύα ιδιοκτησία για τους υπόπτους και είναι πολύ διαφορετικές οι διαδικασίες στα κράτη-μέλη για τα θέματα αυτά και οι αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες. Πολλές φορές μέσα στα κράτη-μέλη τα ίδια πρέπει να υπάρξει εσωτερικός συντονισμός. Πολλές φορές δεν υπάρχει μια ενιαία συντονιστική αρχή στα κράτη-μέλη για να μπορέσει να εξασφαλίσει την εκτέλεση αυτών των ε, αιτήσεων αρρωγής. <clears throat> πολύ συχνά έχουμε καλές περιπτώσεις που δείχνουν την προσθέμενη αξία της ε, Eurojust. Οι Τσέχοι συνάδελφοι είχαν μια έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων και φόρο φοροδιαφυγής, 25 εκατομμύρια <clears throat> ευρώ περίπου. Και είχαν ανακαλύψει ότι ο εμπλεκόμενος λογαριασμός ήταν στην Αυστρία. Μόνο χάρη στην ταχεία διαδικασία συντονισμού μέσω της Eurojust έγινε δυνατόν να υπάρξει κατάσχεση των 25 εκατομμυρίων στον αυστριακό λογαριασμό εγκαίρως, γιατί ο αδικοπράτων, ο οποίος ήταν τότε στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε δώσει την εντολή για μεταφορά αυτών των κονδυλίων. Μετά από δύο ή τρεις ώρες τα λεφτά θα είχαν κάνει πτέρα και επομένως δεν θα τα είχαμε πάρει ποτέ πίσω. Μόνο χάρη στην καλή συνεργασία μεταξύ των Τσέχων και των Αυστριακών συναδέλφων μέσω της Eurojust έγινε δυνατόν να κατασχεθούν αυτά τα χρήματα εγκαίρως. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές στα νομικά και τα δικαστικά συστήματα των χωρών μελών. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πρόβλημα, ιδίως όταν πρόκειται για διαφορά σε σχέση με τον καθορισμό του τι είδου αδίκημα εμπλέκεται κάθε φορά σε μια διαδικασία. Τα φορολογικά αδικήματα μπορεί να είναι διοικητικά αδικήματα ή μπορεί να είναι οικονομικά αδικήματα. Το θέμα είναι αν πρόκειται για παράληψη ή για ηθελημένη ενέργεια. Υπάρχει αμφιβολία γιατί αν πρέπει να εμπλέκονται οι διοικητικέ αρχέ ή οι ιδιοκτικέ αρχέ, όλα αυτά τα στοιχεία απαιτούν λοιπόν κάποιο συντονισμό, ο οποίο είναι και διαμεθοριακού χαρακτήρα. Υπάρχουν επίση ε, δυνητικές συγκρούσεις αρμοδιοτήτων. Ιδίως αν μια έρευνα γίνεται σε μία επικράτεια και θέλουν να ζητήσουν την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων σε ένα άλλο κρατός μέλος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες δυσκολίες γιατί πρέπει να περιμένουν να τελειώσει η πρώτη έρευνα. Επίσης η μεταφορά των ε, ε, αποφάσεων μπορεί να είναι πρόβλημα. Η, επίσης η κατάσχεση προσόδων από, το, από ένα δίκημα, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τους ε, εγκληματίες εκεί που τσούζει, δηλαδή να τους αφαιρέσουμε τα χρήματα. Όλη αυτή η διαδικασία στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες και καθυστερήσεις και αυτό συμβαίνει εάν υπάρχουν τέτοιες διαφορετικές πρόνοιες στα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια τεράστια υπόθεση, τη λεγόμενη κάθετη υπόθεση όπως παρουσιάστηκε στο ερωτηματολόγιο. Αυτό δείχνει τι γίνεται αν υπάρχει πραγματικά συντονισμός. Στη Γερμανία σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε 600 επιστολές αιτήσεων που έπρεπε να σταλούν συντονισμένα και να εφαρμοστούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν το γιγάντιο αυτό έργο το οποίο χρειάζεται να λάβει χώρα. Γι' αυτό το να μπορέσει έγκαιρα να εμπλακεί ένας φορέας όπως η Eurojust είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην περίπτωση των εγγράφων του Παναμά είχαμε μια συνάντηση συντονισμού η οποία ήταν ουσιαστικά η ανακτήρια συνάντηση αυτού του είδους, αυτό το οποίο είδαμε στην περίπτωση αυτή είναι ότι για ένα θέμα τόσο μεγάλης έκτασης και εμβέλειας είναι πολλές φορές δύσκολο και σε επίπεδο και σε ό,τι αφορά την οικονομική και επιμελητιακή του πλευρά να έχουμε συντονισμό. Μία συνάντηση συντονισμού κοστίζει περίπου λίγο, λίγο κάτω από τα 8.000 ευρώ. <clears throat> Στην περίπτωση των συναντήσεων συντονισμού για τα έγγραφα του Πάνωμα, το κόστος ήταν 60.000. <clears throat> Αυτό είναι λοιπόν μια μεγάλη πρόκληση για οποιοδήποτε φορέα. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει λοιπόν είναι και πάλι να εξασφαλίσουμε τον αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων αρχών. Αυτό λοιπόν αξίζει να το σκεφτούμε, <clears throat> να δώσουμε τη δυνατότητα για τις εθνικές ε, αρμόδιες αρχές, τις εισαγγελικές αρχές, να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες που κάποιος από αυτούς έχει αποκομίσει. Αν θέλουμε να συνεργαστούμε με τον Παναμά, Υπάρχουν τρόποι να το επιτύχουμε αυτό. Υπάρχει η διαδικασία αυτή των συναντήσεων <clears throat> συντονισμού αλλά δεν έχουμε κάποιο νομικό εργαλείο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να εξασφαλίζει αυτή την αμοιβαία αρρωγή. Κάποια κράτη-μέλη έχουν κάποια ε, διμερή εργαλεία αυτού του είδους και είναι σε επαφή με τον Πάναμα, αλλά η διπλωματική οδός είναι βραδία και πεπλεγμένη. Αυτό το οποίο χρειάζεται λοιπόν είναι να συνενώσουμε τις ευρωπαϊκές εμπειρίες και ικανότητες μέσα σε αυτή την πλατφόρμα που είναι η Eurojust. Θα το πράξουμε την προηγούμενη εβδομάδα, τις προηγούμενες μέρες αν θέλετε, στείλαμε μια επιστολή στον Παναμά για να τους προσκαλέσουμε σε μια συνάντηση συντονισμού και λαμβάνουμε υπόψη αυτό το οποίο είπε ο Γενικός Εισαγγελέας του Παναμά είπε ότι είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί μας σε δυνατές επίπεδο. Εν κατακλείδη. Είναι κέριος ο ρόλος της Eurojust στον αγώνα κατά του ξεπλήματος χρήματος και της φοροαποφυγής. Μπορούν να υπάρχουν όμως τεχνικά και νομικά προβλήματα που περιπλέκουν αυτή τη διαδικασία, πάντως χωρίς συντονισμό δεν πιστεύω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Και θα έλεγα συνολικά ότι δεν είναι αυτή η χρονική στιγμή, αλλά με υπόψη την περίπτωση του Παναμά και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, να μειώσουμε τη χρηματοδότηση και το επίπεδο στελέχωσης της Eurojust. Το αντίθετο πρέπει να συμβεί, πρέπει να ενισχυθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε και αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε για την ίδια ε, των ε, συζητήσεών μας. Είχαμε συμφωνήσει οι δύο συνεισηγητές να πάρουν το λόγο πρώτοι για να θέσουν ε, ερωτήσεις και να λάβουν και απάντηση σε πέντε λεπτά κάθε φορά. Γι' αυτό θα ήθελα να δώσω τον κύριο Γέπε Κόφοντ, τον λόγο ο οποίος είναι συνεισηγητής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ομιλητές για τις ε, παρουσιάσεις που μας έκαναν και για τις γραπτές ε, απαντήσεις που μας έδωσαν. Να περάσω στην πρώτη ερώτηση πάρα αυτά. Καταρχά, προ τον εκπρόσωπο τη Eurojust, είπατε, αν σωστά θυμάμαι, ότι το 1 τέταρτο του ξεπλήματος ε, χρήματο χρειάζεται διεθνή συντονισμό. Έχετε συγκεκριμένε συστάσει τώρα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζει την οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράμένες δραστηριότητε. Έχετε κάποια σύσταση να μας κάνετε. Τώρα, στο υπόλοιπο πάνελ και στις γραπτές απαντήσεις σας, πολύ αναφερθήκατε στα εμπόδια που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ της αστυνομία και των εθνικών αρχών και το καθεξής. Θα έχει λοιπόν νόημα να δημιουργηθεί ένα τυποποιημένο κεντρικό μητρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι προσβάσιμο από όλα τα κράτη-μέλη, από τις εθνικές αρχές δηλαδή, θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει μια λύσει και την Όλαφ και την Europol ρωτάω και τώρα συγκεκριμένα την Europol. Στις γραπτές απαντήσεις σας νομίζω ότι περιλαμβάνονται πάρα πολύ σημαντικές ε, απαντήσεις και είπατε ότι η Europol έχει λάβει πολύ κατακριματισμένες πληροφορίες από τα κράτη-μέλη και η αστυνομία των κρατών μελών αποφασίζει πότε και αν θα συμμετέχει σε υποθέσει και δεν υπάρχει κάποιο ελάχιστο όριο για τι αποφάσει αυτέ. Πώ μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μέλων, Πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα αποστέλλονται οι σχετικέ πληροφορίε στη Europol, έχετε κάποια συγκεκριμένη σύσταση να μα κάνετε, αντιμετωπίσετε κάποιο εμπόδιο συγκεκριμένα, το οποίο θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μα με κάποιο συγκεκριμένο κράτος μέλος, ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ, συνάδελφε, και να δώσω το λόγο στον κύριο My... Κάμπρι για τις δύο πρώτες ερωτήσεις και μετά στον κύριο Ριοντέ και στον κύριο Κέσλερ. Ο κύριος Μάιερ Κάμπρη. Πέντε λεπτά έχουμε για την ερωτοαπάντηση. Σύνολο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και να μην σχολιάσω για την αναθεώρηση της οδηγίας. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό και γιατί αναφέρθηκα στα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Η φύση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος είναι τέτοια που ως εθνική αρχή δεν μπορούν μάλλον οι εθνικές αρχές να ανταπεξέλθουν σε ό,τι αφορά τον διασυνοριακό χαρακτήρα του εγκλήματος αυτού. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούμε σε μια θέση όπου θα συνεργαζόμαστε, πραγματικά θα συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τρίτα κράτη-μέλη. Σε πολλές περιπτώσεις εμπλέκονται και τριτά αν δεν υπάρχει μια πλατφόρμα συνεργασία, τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Και η πλατφόρμα αυτή, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται και τρίτα μέρη, η εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ διαφορετική όταν μιλάμε, για παράδειγμα, με μία φωνή ως Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση 28 κρατών μελών με κάποιον εξωτερικό εταίρο. Είναι πολύ διαφορετικό από όταν μιλάμε ένας προς έναν. Η πλατφόρμα αυτή υπάρχει ήδη. Είναι η Eurojust. Αυτό όμως που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο η δουλειά αυτή. Θα πρέπει να μπορεί να γίνεται με σωστό τρόπο αυτή η δουλειά. Και αυτό δυστυχώς σημαίνει λεφτά. Σας είπα ποιο είναι το κόστος της ε, συντονιστικής εργασίας. Και συχνά η χρηματοδότηση και ο προπολογισμό για τέτοια θέματα συντονισμού εξατλείται πολύ γρήγορα. Και φυσικά χρειάζεται και προσωπικό η συνεργασία αυτή. Άρα, σας απευθύνω έκκληση. Χρησιμοποιήστε την ήδη φυστάμενη πλατφόρμα για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στις περιπτώσεις αυτές. Σας ευχαριστώ, κύριε Ριοντέ. Thank you for your question. Um, ευχαριστώ για την ερώτησή σας περαιτέρω συνεργασία. Αυτό είναι το αίτημα από πλευρά σας. Κοιτάξτε, η οικονομική άνεση είναι προϋπόθεση και για το οργανωμένο έγκλημα και για τις τρομοκρατικές δραστηριότητες. Είναι λοιπόν ένας σαφής και διαρκής χώρος έρευνας και έχουν γίνει προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Για το μέλλον τώρα θα πρέπει να πείσουμε τις εθνικές υπηρεσίες να συμμερίζονται ε, τα στοιχεία τους και τις εμπειρίες τους με την Europol. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει περισσότερη συνεργασία και περισσότεροι συμμετέχοντες στη συνεργασία αυτή για να δούμε ακριβώς τι γίνεται γύρω από τις ύποπτες συναλλαγές ε, της ε, τραπεζικές. Εμείς ξεκινήσαμε ε, τον Ιανουάριο με την ενσωμάτωση των ρυθμίσεων αυτών στις ε, διάφορες υπηρεσίες και τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες και στην Europol. Αν γίνει αυτό τότε η συνεργασία σαφώς θα ε, έχει ανέλθει σε επίπεδα όταν υπάρχουν κάποιες νομικές δεσμεύσεις και νομικές τροχοπέδες για την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις διαφορετικές υπηρεσίες, είναι σαφές ότι σήμερα είναι πιο απαραίτητο από ποτέ τα FIU να μπορούν να ανταλλάσσουν τις υπηρεσίες και όχι μόνο μεταξύ κατασταλτικών υπηρεσιών, αλλά και τελωνιακών υπηρεσιών, χωρίς περιορισμούς από εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις. νομίζω ότι η συνεργασία με τη Europol μπορεί να λειτουργήσει συγκεντρωτικά και συντονιστικά. 30 seconds for... Ευχαριστώ. 30 δευτερόλεπτα για το Ζωβάνι. Τι... τι... Regulation on, the directive, actually on the money. Η, για την οδηγία για το money laundering. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη μας και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουλίου του 2016 έτσι ώστε όλοι τα FIU να είναι σε θέση να συμβουλεύονται τις τράπεζες δεδομένων των μεμονωμένων χωρών μελών το βήμα το επιπλέον, το οποίο προς το παρόν δεν έχει προταθεί ε, επίσημα, αλλά μπορεί να υπεστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν παράδειγμα, θα πρέπει οι τράπεζες αυτές δεδομένων να είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες σε όλες τις ελεγκτικές αρχές, εποπτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο δεύτερο πάνελ μάλλον στο δεύτερο συνεισηγητή, τον κύριο Γετσέκ, δεν είναι παρόν, αλλά έχει, θα το αντικαταστήσει ο κύριος Λουί Μισελ. Δυστυχώς ο κύριος Γετσέκ δεν μπορεί να είναι παρόν, λέει ο κύριος Μισελ. Πρώτη σκέψη προς τους τρεις παρεμβαίνοντες. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Μιλήσατε πολύ για την συνεργασία μεταξύ σας και γενικά για τον συντονισμό και τη συνεργασία. Βέβαια υπάρχει το πρόβλημα ότι υπάρχει έλλειψη ε, αποδοτικότητα σε αυτή τη συνεργασία η οποία απαιτεί πάρα πολλή εργασία. Και δεύτερον στέκομαι στην παρέμβαση του κύριου Κέσλερ, ο οποίος είπε κάτι ενδιαφέρον. Μίλησε για ένα μητρό των τραπεζικών λογαριασμών. Ένα ερώτημα που θέλω να σας θέσω κύριε Κέσλερ, γιατί το ακούω αυτό πολλές φορές, η νομοθεσία <clears throat> για την προστασία της προσωπικής ζωής εμποδίσουμε το έργο έρευνά σα και το έργο συντονισμού. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό, γιατί πολλές φορές κάνουμε μία προσπάθεια είναι μια προσπάθεια να εμποδίζεται η παροχή στοιχείων λόγω της προστασίας δεδομένων. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Και δεύτερον, πάντα κάνουμε τη διάκριση μεταξύ λεύκανσης χρημάτων ε, απάτης, φοροδια, φοροδιαφυγής, απάτης και της λεγόμενης βελτιστοποίησης στα φορολογικά θέματα. Αυτά οι διαφορετικοί ορισμοί πολλές φορές διαφορούν και δημιουργούν και κάποια σύγχυση η οποία αποδυναμώνει και το δικό σας ρόλο και το έργο μας. Θα ήθελα λοιπόν και θέτω το ερώτημα στους, σε όλα τα μέλη του πάνελ μήπως πρέπει να υπάρξει κάποιος προβληματισμός μήπως θα μπορέσουμε κάποια μέρα να έχουμε μια κοινή, ένα κοινό ορισμό όλων αυτών των ενιών, οι οποίες επικαλύπτονται σε κάποιο βαθμό. Γιατί τώρα μεταξύ φορολογικής ευελτιστοποίησης και της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα να τα ξεκαθαρίσουμε, αλλά θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη σαφήνεια. Και ένα ακόμα ερώτημα. Έχω ακόμα χρόνο, λέει, όχι. Εντάξει, θα επανέλθω αργότερα, λέει ο κύριος Μισελ. Σας ευχαριστώ κύριε Μισελ. Κύριε Κέσλερ, ε, ετέθησε ένα ερώτημα. Η προστασία των ε, δεδομένων των προσωπικών είναι θέμα φυσικά Προστασία των ιδιωτικών δεδομένων, εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία το θέμα είναι ότι οι νομοθέτες μερικές φορές πρέπει να συντενίζονται μεταξύ τους, γιατί μερικές φορές ε, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην προστασία των δεδομένων από τη μία και τις προβλέψεις για τις διαρευνητικές ανακριτικές διαδικασίες από την άλλη και δημιουργείται μια κάποια σύγχυση που για μας αποτελεί πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποστηρίζουμε πλήρως, αλλά αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι εμείς προσπαθούμε να λειτουργήσουμε και σε επίπεδο ε, διερευνητικό και σε επίπεδο ε, θεματοφύλακα, αν θέλετε, των νομοθεσικών ρυθμίσεων, αλλά πολλές φορές αυτό μας φέρνει σε αδιέξοδο. Το θέμα λοιπόν των προσωπικών δεδομένων δεν είναι πρόβλημα για μας, απλά πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρες οι νομοθετικές ρυθμίσεις. Για το τελευταίο τμήμα της παρέμβασής σας, κύριε Μισελ, εγώ έχω την αίσθηση ότι μπορώ να εκφραστώ υπέρ μιας μη πολύ διασπασμένης αντιμετώπισης ε, του νομοθέτη πάνω στην ε, προστασία των δεδομένων. <clears throat> Αλλά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι κάτι παραπάνω. Και το ξέρω ότι το ξέρετε, το ξέπλυμα ε, υπάρχει σαν αποτέλεσμα μιας άλλης ποινικά κολάσιμης δραστηριότητας Οπότε είναι λίγο περίεργο το να μπορούμε να διερευνούμε το βρώμικο χρήμα χωρίς να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε τα ίδια δεδομένα για την προηγούμενη ε, ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά. Αυτό που απαιτείται λοιπόν είναι μια ενιαιοποιημένη, αν θέλετε, νομοθετική αντίληψη. Ευχαριστώ πολύ, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος τώρα θέλει το λόγο, οπότε τώρα Έχουμε καλύψει τα πέντε λεπτά. Ο κύριος Όθμαρ Κάρας έχει το λόγο, παρακαλώ, για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, είναι απλό και σύντομο το ερώτημά μου προς όλα τα μέλη του πάνελ. Υπάρχει η πλατφόρμα των δημοσιογράφων, το Διεθνές Consortium των Ερευνητικών Δημοσιογράφων το ερώτημά μου είναι με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό συνεργάζεστε με αυτή την πλατφόρμα των δημοσιογράφων. Έχετε ζητήσει για κάποια έγγραφα από τους δημοσιογράφους, έχετε πάρει κάποια σχετικά έγγραφα, έχετε την εντύπωση ότι θα σας δοθούν τέτοια έγγραφα από το Consortium. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Κύριε Μάιερ Κάμπρι. είναι, όπως σας είπα, δεν είναι μέσα στα καθήκοντα της Eurojust να κάνει έρευνες. Απλώς εμείς συντονίζουμε. Επομένως εμείς δεν έχουμε συνεργασία με αυτή την πλατφόρμα, εκτός από τις περιπτώσεις που πρέπει να παρέμβουν οι εθνικές εισαγγελικές αρχές. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό άμεσα από τη Eurojust. Κύριε Ριοντέ, η Europol Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα άμεση επαφή με το consortium των δημοσιογράφων. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και χρειαζόμαστε την αρρωγή των κρατών μελών για να πάρουμε δεδομένα. Εμεί μπορούμε να έχουμε επαφή μόνο στα ε, δεδομένα τα οποία μας δίνουν τα κράτη-μέλη, που είναι η μόνη πάροχη δεδομένα. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από το consortium αυτό των ε, δημοσιογράφων. Εμείς αντίθετα με τους συναδέλφους μου εγώ εκπροσωπώ ένα φορέα ο οποίος είναι ερευνητικού χαρακτήρα και γι' αυτό ήρθαμε σε επαφή και με τους δημοσιογράφους. Εμείς λοιπόν λειτουργήσαμε επί τη βάση των δημόσια διαθέσιμων στοιχείων. Πρόκειται για στοιχεία που ήταν δημόσια και μετά ήρθαμε σε επαφή με τους δημοσιογράφους και είχαμε κάποιο εκπρόσωπο ο οποίος ήρθε ενώπιον της Όλαφ και ζητήσαμε να έχουμε και τα υπόλοιπα έγγραφα τα οποία δεν έχουν γίνει απόλυτα, δεν έχουν γίνει δημόσια και τα οποία θα ήταν χρήσιμα και για τις έρευνες μας. Η απάντηση μέχρι στιγμής ήταν όχι. Και ο κύριος λόγος για κάτι τέτοιο, φυσικά δεν έχουμε τη δυνατότητα να ε, απαιτήσουμε τα έγγραφα αυτά, πάντως έχουν τη δυνατότητα να το ζητήσουμε, να τα πάρουμε. Ο κύριος λόγος για την άρνηση από το, την Consortium είναι γιατί αν αποκαλύψουν όλα αυτά τα έγγραφα, αυτό μπορεί να αποκαλύψει και κάποιες πηγές και να θέσει τις πηγές σε κάποιο κίνδυνο. Και φυσικά εμείς δεν πρόκειται να πληρώσουμε κάποιον όπως έκαναν οι φορολογικές αρχές της Δανίας για να πάρουμε DVD ή οποιαδήποτε άλλη πηγή στοιχείων. Λοιπόν, πήραμε και στην πρώτη ακρόση που κάναμε με τους δημοσιογράφους ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτούς η προστασία των πηγών τους και σε αυτήν οφείλεται και η επιφυλακτικότητά τους στο να δώσουμε δεδομένο. Ο για συντοματικό ερώτημα. Γνωρίζω το πρόβλημα αυτό, είναι σοβαρό, αλλά ξέρουμε ότι δεν έχουν δοθεί όλα τα έγγραφα, δεν ξέρουμε ότι, ξέρουμε ότι αυτό δεν έχει γίνει, αλλά και ο πρώτος από τους ομιλητές μας είπε ότι οι εθνικές εισαγγελικές αρχές μπορούν να δώσουν στοιχεία. Πώς λοιπόν λειτουργεί αυτή η συνεργασία σας με τις εθνικές εισαγγελικές αρχές και με τις ερευνητικές αρχές στα κράτη-μέλη και μπορείτε να ελέγξετε αν δόθηκαν από αυτούς τέτοιου είδους στοιχεία ή όχι. Παρακαλώ μια σύντομη απάντηση. Να σας ε, παραπέμψω στην ε, παρουσίαση των ε, εθνικών αρχών, εισαγγελικών και αστυνομικών, οι οποίες μπορούν να σας δώσουν περισσότερα στοιχεία, λέει ο κύριος Κάμπρη. So far we haven't received much. Ως τώρα Έχουμε λάβει κάποια στοιχεία, μας πήρε κάποιο χρόνο η ανάλυση των δεδομένων αυτών και να καταλήξουμε στις 3.400 hit. Ε, και αυτά τα πακέτα χωρών λοιπόν θα αποσταλούν αυτή την εβδομάδα και θα περιμένουμε τις απαντήσεις και τα δεδομένα τα οποία θα μας δώσουν τα κράτη-μέλη. Βρισκόμαστε λοιπόν το μέσο της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ λέει, λέει ο Πέτρος, οι σοσιαλδημοκράτες, ο κ. Ράμο Ανατόντο. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να θέσω το ερώτημα για το πλαίσιο σχέσεων που υπάρχει μεταξύ των φορέων σας με τις υπηρεσίες και τις διοικητικές δομές ε, των ε, φορολογικών αρχών κάθε χώρας, γιατί συζητάμε και ο κύριος Ριοντέ το έχει ε, εξήγηση αυτό. <clears throat> Υπάρχει μια κάποια μομφή έμεση η οποία έχει δημιουργηθεί έναντι του consortium των δημοσιογράφων για το γεγονός ότι είναι ορισμένες πληροφορίες αλλά όχι άλλες. Μα χάρη σε αυτούς υπάρχουν τα έγγραφα του Παναμά, χάρη στους δημοσιογράφους. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να συζητάμε αν αυτοί πρέπει να δώσουν περισσότερε πληροφορίε, λιγότερε πληροφορίε, όταν αυτοί έκρουσαν τον κόνδωνα του κινδύνου για αυτό το σοβαρό θέμα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέλω να θέσω ιδίω προ την Ευρωπόλ. Μήπω έπρεπε να είναι τα κράτη-μέλη αυτά τα οποία θα έπρεπε να σα δίνουν τι πληροφορίε που χρειάζεστε. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μα πούν τι ακριβώ είναι αυτό το οποίο χρειάζεστε ω Ευρωπόλ. Δεν θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Δεύτερο θέμα προ την Eurojust Υπάρχουν κάποιες χώρες που ζήτησαν μέσα στη Eurojust να γίνει έρευνα για τα έγγραφα του Παναμά. Δηλαδή, δεδομένου ότι το έργο σας είναι έργο συντονισμού των εθνικών εισαγγελικών αρχών, υπήρξε κάποια εθνική αρχή εισαγγελική που ζήτησε από τη Eurojust να κάνει κάτι για τα έγγραφα του Παναμά. Και τρίτο ερώτημα. Πώς συνδέεται ο δικός σας φορέας με τα αστυνομικά και δημοσιονομικού χαρακτήρα φορολογικές αρχές των κρατών μελών τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ακόμα και τράπεζες όταν υπάρχει ξέπλυμα χρημάτων ή οικονομικό έγκλημα. Ποιε είναι οι σχέσει με αυτέ τι αρχέ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ και ποιο θα ξεκινήσει, ο κύριος Βιοντέ. Σε ό,τι αφορά το ICIG, δεν υπάρχει κάποια έκθεση από, την... από το σώμα αυτό ως μια υπηρεσία όμως που παρέχει υπηρεσίες προς τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα η τέταρτη οδηγία κατά του ξεπλήματος βραμικού χρήματος και σε ό,τι αφορά τα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών. Θα θέλαμε να υπάρχει δυνατότητα να μας δώσουν τα κράτη-μέλη τις πληροφορίες αυτές. Ασφαλώς με χαρά θα ερευνήσουμε οποτεδήποτε υπάρχει κάποια, κάποια δίκημο. Αυτό λοιπόν θα το διαβιβάσουμε στα κρατημέλη. Ο κύριος ε, Μάιρ Κάμπρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τα δύο αυτά ερωτήματα προς την κύριο Και όντως, μας ατήθηκε να υποστηρίξουμε τις εθνικές έρευνες και εγώ είμαι εδώ ως εθνικό μέλος της Γερμανίας. Γιατί το πρώτο αίτημα προήλθε από τη Γερμανία. Έτσι λοιπόν είναι πλάκη η Eurojust. Και έτσι εμπλέκονται και τα υπολοιπα κρατημέλη τη Ένωση. Η συνεργασία με τη ΣΥΠΑ. Η Eurojust έχει συμφωνία συνεργασία με τη ΣΥΠΑ. Και η ΕΠΑ μετά την Ελβετία και την Νορβηγία είναι οι μοναδικέ τρει χώρε που έχουν ξεκινήσει μια τέτοια συνεργασία με τη Eurojust και η συνεργασία λοιπόν βασίζεται στη συμφωνία αυτή και ουσιαστικά είναι σαν να είναι κράτο Είναι εξαιρετικά η συνεργασία με τις τρεις αυτές χώρες, λοιπόν. Ο κύριος Κέσλερ. Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι το κράτος μέλος ή εμείς αυτοί που θα βρουν τα 11 εκατομμύρια έγγραφα τα οποία είναι στα χέρια των δημοσιογράφων. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν έχει την εξουσία να τα κατάσχει. Σίγουρα όχι όλα αυτά, αλλά ούτε και οι εθνικέ αρχέ. Δεν έχουν αρμοδιότητα. Δεν έχουν και το ένωμα μέσα. Για να συλλέξουν όλα αυτά τα στοιχεία, όλα αυτά τα έγγραφα, τα οποία ενδεχομένω να αποτελούν τεκμήρια για οποιοδήποτε έγκλημα, τίθεται θέμα νομική αρμοδιότητας. Δεν ξέρουμε και πού είναι αυτά τα έγγραφα. Άρα, όλοι ξεκινήσαμε έρευνες, γιατί αυτοί αποφάσισαν να διαθέσουν τμήμα των εγγράφων αυτών. Άρα, το μόνο που μπορούμε να δούμε ως ε, λύση είναι η περαιτέρω συνεργασία μαζί τους. Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς, αλλά να συνεργαστούμε προκειμένου να σχηματίσουμε μια πιο δίκαιη και ολοκληρωμένη εικόνα. Σας ευχαριστώ, ο Πρόεδρος. Ακριβώς πέντε λεπτά. Επόμενη ομιλήτρια από το ECR. Kiitos puheenjohtajalle ja asiantuntijoille. Ehdotus uudeksi rahan... Σχετικά με την εφαρμογή της νέας οδηγίας. Η νέα οδηγία σαφώς περιλαμβάνει πολλές ε, θετικές πρωτοβουλίες οι οποίες ε, καθιστούν πιο διαφανή τα στοιχεία. Βέβαια οι ρυθμίσεις έχουν ορισμένα αρνητικά στοιχεία. Δυσκολίες, σαν παράδειγμα, στην έβρεση του πραγματικού ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης. Και επίσης ε, φορολογική παράδειση, όχι μόνο Παναμά, αλλά και άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτά τα παραθυράκια λοιπόν πώς θα καλυφθούν. Πώς θα μπορέσουμε ε, να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά τα στοιχεία και τι σημαίνει αυτό για την καταπολέμηση σε διεθνές επίπεδο ε, στον τομέα ε, του βρώμικου χρήματος. Μια δεύτερη ερώτηση εσείς ε, όταν ε, ε, διασταυρώνετε τα στοιχεία σας αναφέρεστε στην έβρεση συγκεκριμένων προσώπων και υπηρεσιών που εργάζονται στα θεσμικά όργανα. Γιατί ύψους πιθανές ζημίες μιλάμε σε αυτή την περίπτωση. Να ξεκινήσω, λέει ο κ. Κέσλερ, από τη δεύτερη ερώτηση. Κοιτάξτε, σας είπα ότι τα αποτελέσματα της αναλυτικής προσπάθειας την οποία κάναμε μέχρι τώρα δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ε, ε, τροτά στρατηγικής φύσεως σημεία σε επίπεδο κοινοτικού προσωπικού ή σε επίπεδο θεσμικών οργάνων. Σας είπα ότι βρήκαμε ε, ταυτίσεις μόνο σε 17 περιπτώσεις από 40 ή τόσες χιλιάδες. Καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ περιορισμένος και μετά από ε, τις συγκεκριμένες διαδικασίες επιλογές εμείς ξεκινήσαμε μόνο τέσσερις έρευνες γιατί οι υπόλοιπε περιπτώσεις ήδη αναφέρονταν σε έρευνες οι οποίες είτε έχουν κλείσει είτε διεξάγονται ακόμα και τώρα. Οκτώ λοιπόν μόνο ταυτίσεις περιελάμβαναν νέα στοιχεία και από τις οκτώ μόνο οι τέσσερις οδήγησαν σε νέες έρευνες μετά από σε βάθος ανάλυση των στοιχείων. Ενώ οι άλλες ήταν συνωνυμίες κτλ. Λοιπόν, τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ε, τροτά στοιχεία συστημικά. Αντίθετα υπάρχει ένα υψηλότατο επίπεδο καθαρότητας θα έλεγα στα ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα και στο προσωπικό τους. και από τις τέσσερις περιπτώσεις που ερευνούμε μόνο η μία αφορά ε, κοινοτικό υπάλληλο, δηλαδή ένα πολύ μα πολύ μικρό ποσοστό. Απαντήσεις από τους... Ε, χρειάζεστε να απαντήσετε, όχι? Εντάξει. Επειδή έχουμε καθυστερήσει λιγάκι, μπορούμε να περάσουμε στην κυρία Παπακατσόντα από την Άλντετ. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν να σας συγχαρώ όλους για την... και να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι κάτι γίνεται, κάτι μαθαίνουμε και όλες οι προτάσεις οι οποίες έχουν παρουσιαστεί από εσά είναι πράγματα που εμείς θα τα λάβουμε υπόψη για το έργο μας. Τώρα το ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω στον κύριο Ριοντέ. Ποια κάτι μελη ζήτησαν τη συνεργασία της Όλαφ στη Γυροπόλ, συγγνώμη για τη διαρροή των εγγράφων του Παναμά και κατά πόσο γνωρίζετε αν θα δημιουργηθεί ένα κέντρο εμπειρογνωμοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά βάσει του άρθρου 4.1 του κανονισμού της Ευρωπόλ που θα τεθεί σε λειτουργία του χρόνου. Μας μιλήσατε για υψηλό επίπεδο τώρα ακαιρεότητας για το προσωπικό και τους εμπλεκομένους. Αυτό μας χαροποιεί και τους επιτρόπους που είπατε, αλλά υπάρχει το θέμα των ε, ε, άμεσων συγγενών των επιτρόπων. Έχετε προβλέψει, επειδή έχει βγει κάπως ε, φιλτραρισμένο το έγγραφο του Παναμά, επειδή ένα από αυτό έχει να κάνει με τη σύζυγο του κυρίου Κανιέτε, του Επιτρόπου. Θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η άποψή σας για αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Ο κύριος Κέσλερ, ποιος θα ξεκινήσει ή η Τα Θα μπορούσατε παρακαλώ να επαναλάβετε την ερώτηση για το εξειδικευμένο αυτό κέντρο. Συγγνώμη, λέει η κυρία η Μάιτε. Στον κανονισμό της Europol που θα τεθεί σε εφαρμογή και θα ενισχύει τις δυνατότητες δράσης της Europol, εμφανίζεται η δυνατότητα στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ε, υπό παράγραφος L λατινική να υπάρξει ένα κέντρο παροχής συμβουλών ειδικευμένο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Θα θέλαμε να ξέρουμε αν αυτό το εργαλείο προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία θα ήταν πολύ χρήσιμο για τον καλύτερο συντονισμό στα θέματα αυτά τα οποία αναφέρατε και θέλω και πάλι να σας συγχαρώ για αυτά που μας είπατε. Εντάξει, παρακαλώ. Στην παρούσα φάση γύρω από όλα αναμένει την εφαρμογή της τέταρτης ε, οδηγίας ε, για την ε, καταπολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου κέντρου ε, χρήματος για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πόρους μας και επικεντρωνόμαστε κυρίως στην νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Α, θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Για το θέμα για την ΟΛΑΦ. Ένα από τα ονόματα τα οποία ψάξαμε στο σύστημα στη βάση δεδομένων είναι ονόματα εταιριών και ονόματα αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβασιούχου. Όχι τα ονόματα μελών της οικογένειας, ε, κύριε Μισελ, για θέματα προστασίας των δεδομένων κτλ. Γιατί πραγματικά θα ήταν ένα τεράστιο ψάρεμα αυτή η διαδικασία, αυτή η άσκηση. Άρα δεν λάβαμε ε, τέτοια hit για μέλη της οικογένειας, μόνο για άτομα τα οποία έχουν εργαστεί στα θεσμικά όργανα. Ωστόσο, ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο στη φούσκα αυτή των Βρυξελών και ξέρουμε διαβάζοντας τα τις εφημερίδες, όχι απαραίτητα τις ισπανικές, ότι υπάρχουν και μέλη οικογένειας αξιωματούχων υπαλλήλων που ενδεχομένω να μας ενδιαφέρουν. Και πρέπει να σας πούμε ότι η πολιτική μας είναι ότι δεν δημοσιεύουμε τα ονόματα των όσων ερευνούμε. Ελπίζω να με νοήσετε. Σας ευχαριστώ. Από την ΚΟΕ τώρα, Μιγκουέλ Βιέγκας. Eh, Είχα κάποια ερωτήματα. Εμείς ε, Συμμεριζόμαστε την ανάγκη να υπάρξει βελτίωση των κανονισμών, την βελτίωση των εργαλείων έρευνας, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που βλέπω, αυτό το οποίο δεν μπορούμε <clears throat> να παραγνωρίσουμε είναι δύο βασικά εμπόδια σε αυτόν τον αγώνα. Ο πρώτο, το πρώτο εμπόδιο έχει το, να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος βασίζεται πάρα πολύ στην πρέπουσα ε, στην πρέψου ευσυνειδησία και επομένως ε, δεν δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει η αποκάλυψη υπό, υπόπτων συναλλαγών και δεύτερον το γεγονός ότι δεν έχουμε την υποστήριξη από επιλογνωμόνες. Πώς λοιπόν μπορείτε εσείς να δείτε οι κυβερνήσεις να παρέμβουν με πιο στεναρό τρόπο ώστε να υποχρεώσουν τους ε, χρηματοπιστωτικούς φορείς και τους άλλους φορείς που εμπλέκονται στην λεύκαση κεφαλαίων να δίδουν τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Γιατί αυτό το οποίο διακρίνω μέσα από τις απαντήσεις που πήραμε είναι ότι δεν κυκλοφορεί η πληροφορία. Είτε σε ό,τι πρόκειται για ύποπτε συναλλαγέ, είτε για του τελικού δικαιούχου αυτών των συναλλαγών. Πολύ λίγε χώρε κάνουν κάτι για τα θέματα αυτά και και ένα δεύτερο θέμα που έχει να κάνει, όχι με τους εμπειρογνώμου, συγγνώμη, με τους φορολογικούς παραδείσους, είναι ότι μία από τις βασικέ ανάγκες για την παρέμβαση των κυβερνήσεων είναι με το να απειλήσουν ότι θα ασκήσουν κυρώσει εναντίον των φορέων που εργάζονται με φορολογικούς, συνεργάζονται με φορολογικού παραδείσου. Αυτό όμω σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα κατάλογο φορολογικών παραδείσων ο κατάλογος αυτός όμως βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγμάτευση, αφορά μονάχα Τρίτε χώρες, δεν περιλαμβάνει χώρες καθόλου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει κριτήρια που να επιτρέψουν χώρες όπου είναι μηδενική η φορολογία να ενταχθούν σε αυτό το κατάλογο. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η άποψη του πάνελ για αυτέ τι εργασίε που λαμβάνουν χώρα σε αυτό το τόσο ευαίσθητο τομέα. Για τον ε, ε, μαύρο κατάλογο για τη μαύρη λίστα υπάρχουν προτάσεις στην ΕΚΟΦΗΝ σε σχέση με τον κατάλογο των φορολογικών παραδείσων. Θέλετε να απαντήσετε, ο κύριος Μάιερ Κάμπλη. Να αναφέρω μία πτυχή και να απαντήσω στο θέμα της συνεργασίας με τα κράτη γενικότερα. Αυτό ασφαλώς είναι πολύ διαφορετικό από αυτά που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. εδώ σε ό,τι αφορά θέματα ποινικού δικαίου και αιτήματα νομικής αρρωγής. Είναι πολύ πιο δύσκολο να χρησιμοποιούμε τη διπλωματική οδό, την οποία χρησιμοποιεί ένα μόνο κράτος μέλος. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ αργά και πάρα πολύ βρατικίνητα και δύσκολα. Από πλευρά μου λοιπόν έχω να πω ότι ω οργάνωση δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Αν υπάρξει μια συνθήκη, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο αυτόματα, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα. Θα υπάρχουν τα σωστά θεμέλια. Αλλά στην παρούσα φάση είναι δύσκολα τα πράγματα και ως εκ τούτου χρειάζεται ένα σώμα το οποίο τουλάχιστον να μπορέσει να αξιοποιεί τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς πόρους. και να αντιμετωπίζει το θέμα των τρίτων χωρών. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Αυτό θα μπορούσε λοιπόν να συμπεριληφθεί ω πόρισμα τη συζήτησή μα. Θα ήθελα να συνεχίσω. Και αυτό γιατί έχουμε και χρονικού περιορισμού. Η κυρία Μόλι Κόρτ κάτω από του Πράσινου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρο. Ευχαριστώ και του τρει ομιλητέ που βρίσκονται εδώ μαζί μα σήμερα για να απαντήσουν τι ερωτήσει μα. Εγώ έχω να ρωτήσω θέματα προ την Europol. Να θέσω ερωτήσει προ την Europol λάβαμε κάποιες πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες μιας χώρας που λέει ότι δεν λάβανε ούτε μία καταγγελία που να σχετίζεται με τα έγγραφα του Παναμά. Πώς γίνεται αυτό, πιστεύετε ότι ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά αυτές τις οικονομικές, μυστικές υπηρεσίες και πώς λαμβάνουν ή δεν λαμβάνουν πληροφορίες σε εθνικό επίπεδο. Αν υπάρχει πρόβλημα, πώς θα το επιλύσουμε. Κατά δεύτερον, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία από κοινού ε, αντιπροσωπεύουν το 70% των υπόπτων συναλλαγών. ω Βρετανή λοιπόν εκπρόσωπος εδώ πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι που λαμβάνουν πολλές ε, πληροφορίες η μυστική υπηρεσία για το οικονομικό έγκλημα της υπηρεσίας της χώρας μου. Γιατί όμως ε, άλλες χώρες όπως η Κύπρος, η Μάλτα δεν λαμβάνουν αντίστοιχο αριθμό καταγγελιών. Τι γίνεται στις χώρες αυτές. Και τέλος, από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου, δεδομένου και του Brexit, και δυστυχώς κάθε μέρα στην χώρα μου πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το Brexit. Ανησυχώ γιατί φοβάμαι ότι ενδεχομένω αυτό να το χρησιμοποιήσουν όσοι θέλουν να αποφύγουν από πλευράς εταιριών την καταβολή ΦΠΑ. Τι επίπεδο λοιπόν ανταλλαγής πληροφοριών θα μπορέσει να διατηρηθεί μετά την αποχώρηση του Ιμνου Βασιλείου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί τα έγγραφα του Πάναμα αποκάλυψαν ότι πάνω από τις μισές σχετικές εμπλεκόμενες ε, εταιρείε είναι στην Ηνωμένο Βασίλειο. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε μετά τον Brexit σήμερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ποιος θέλει να πάρει το λόγο για να απαντήσει. Ο κ. Ριόντε. Σε ό,τι αφορά την πρώτη σας ερώτηση. Όταν το FIU δεν έλαβε κάτι, μάλλον επειδή δεν λάβαμε σχετικές πληροφορίες, θα αποστείλουμε τα πακέτα των χωρών στις διάφορες εθνικές ε, υπηρεσίες. Είναι ευθύνη μετά των κρατών μελών να τα μοιράσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες ε, που τις αφορούν. Σε ό,τι αφορά το Λουξεμβούργο και την Κύπρο και το ερώτημα που θέσατε, δεν έχω κάποια απάντηση να δώσω εγώ ε, παρέχω στην υπηρεσία σας, στην επιτροπή σας μάλλον, τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τις εκάστοτε χώρες. Μία προσθήκη? Όχι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Επόμενος από το EFTD, ο κύριος Μαρκοβάλη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με χαρά βλέπω ότι μετά από το σκάνδαλο των εγγράφων του Παναμά έχουν ξεκινήσει τέσσερις έρευνες. Καταλαβαίνω όλο τώρα τους λόγους για τους οποίους δεν μπορείτε να μας δώσετε λεπτομερικές πληροφορίες για τις εξελίξει έρευνες. Θα μπορούσατε μας να μας πείτε αν είναι σε καλό σημείο αυτές οι έρευνες, αν θα χρειαστεί πολύς χρόνος ή όχι για αυτές τις ε, έρευνες και αν μπορείτε να μας δώσετε και κάποια στατιστικά στοιχεία για να μας εξηγήσετε αν στις έρευνες αυτές εμπλέκονται μέλη του Κοινοβουλίου, μέλη του προσωπικού, μέλη της Κομισιόν κτλ. ή προσωπικό της Κομισιόν κτλ. και εν γέννη για τους άλλους ε, φορείς θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία έχουν συνεργαστεί περισσότερο ή λιγότερο. Αυτό βέβαια το παίρνουμε, τις φορές αυτές παίρνουμε περισσότερο όταν συζητάμε με, στα πλαίσια της Επιτροπής ΤΑΞ. Και επίσης για το κατά πόσο εφαρμόζεται ο κώδικας συμπεριφοράς. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν ε, στην αρχή δώσει μεγάλη έμφαση στην αντιμετώπιση της ε, φοροδιαφυγής ενώ στη συνέχεια έχουν απομονωθεί μέσα στα πλαίσια των επιτροπών που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Φαίνεται να είναι μονάχα μερικές χώρες που έχουν επιθετική συμπεριφορά για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Πρώτα σε εσάς απευθυντική ερώτηση. Δεν... νομίζω ότι μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για τις τέσσερις έρευνες οι οποίες αυτή τη στιγμή εξελίσσονται. Είπα, δεν είναι καμία πάνω σε, προσωπικά, σε μέλη προσωπικού του και των κοινοτικών οργάνων. Θα ήθελα επίσης να πω το ότι το γεγονός ότι ένα μέλος ή ένας υπάλληλος εμπλέκεται, αναφέρεται στα Panama Papers ή έχει ένα δικό του λογαριασμό ή μία εταιρεία κτλ. Αυτό από μόνο του μπορεί να μην είναι ε, ποινικά κάτι που πρέπει να ερευνηθεί. Το θέμα είναι οι οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με την θέση που έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχουν δηλωθεί, καταχωρηθεί, αδειοδοτηθεί και σε αυτή την περίπτωση ε, εξετάζεται αν υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος ή και να μην υπάρχει ή μπορεί να είναι κάποιες οικονομικές δραστηριότητες αυστηρά προσωπικές και αναζητείτε εκεί αν μπλέκετε σε απάτη, σε καταχρηστική ε, συναλλαγή κτλ. Αυτό είναι αυτό το οποίο α, μας απασχολεί, αλλά όπως σας είπα οι διαδικασίες αυτές δεν κρατάνε πάρα πολύ το θέμα είναι ότι αν εμείς είχαμε πρόσβαση στα 11 εκατομμύρια εγγράφων τα οποία δεν είναι δημοσιεύσιμα, αυτό θα μας βοηθούσε πολύ περισσότερο και αυτό θα μας επέτρεπε ε, πράγματι να ξέρουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Ευχαριστώ ευχαριστώ κύριε Σκάπρη για να μας απαντήσει επίσης. Ναι. Και από δική μου πλευρά επιτρέψτε μου να πω το εξή ότι η συνεργασία των κρατών μελών ήταν εξαιρετική. Ε, πρόκειται για το μεγαλύτερο συντονιστικό τέτοιο εγχείρημα, μεγαλύτερη τέτοια συντονιστική συνάντηση σε επίπεδο Eurojust. Το ίδιο ισχύει και για τη Γεροπόλου. Για, για την επόμενη συνάντηση, συντονιστική συνάντηση, θα έχουμε και εκπρόσωπο της όλα, φαντάζομαι. Άρα, πρέπει να σας πω ότι συνολικά είμαι πολύ ικανοποιημένο σε ό,τι αφορά την συμμετοχή των κρατών μελών στις ποινικέ αυτές δραστηριότητε. Σας ευχαριστώ. Δεύτερος γύρος τώρα. για το ΕΛΚ. Μία ερώτηση έχω να σας κάνω. Με τα τρία, από τις τρεις υπηρεσίες μπορείτε να μας πεις ποια κράτη-μέλη είναι α, εκείνα που δεν συνεργάζονται, που μας δυσκολεύουν. Μας είπατε ότι έχετε αναγκαστεί να στείλετε 600 επιστολές σε μία περίπτωση. Πού λοιπόν θα πρέπει να υποκινήσουμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν καλύτερα. Ο κύριο Τριοντέ, ποιος θα ξεκινήσει, ο κύριος Καμπρί. Um, Θα ήθελα να πω το εξή. Αυτές οι 600 επιστολές τις ανέφερα για να σας δείξω το μέγεθος του προβλήματος. Αλλά δεν σημαίνει ότι είχαμε 600 προβληματικές περιπτώσεις, γιατί τα πράγματα πήγαν πολύ καλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακριβώς επειδή υπήρχε πρώτερο συντονισμό και συνεργασία. Η έκταση, ωστόσο, αποτελεί ένα πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν παίρνουμε. Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό των εγγράφων του Παναμά, βρισκόμαστε στην αρχή τη διαδικασία τα πράγματα πάνε καλά. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο κράτο μέλο που μας δυσκολεύει στην παρούσα φάση. Μάλιστα. Μήπως μετά από αυτό που είπε ο κύριο Βάλη, μήπω είναι τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία παρουσιάζουν τα πιο πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά του φορολογικού παραδείσους ή δεν διαπιστώνεται κάτι τέτοιο. Δεν θα ήθελα να αναφέρω ονόματα, αλλά να ξέρουμε. Σχετικά με την Όλαφ, εμείς ε, εντάξαμε τις δραστηριότητες μας στην εντολή που έχουμε από τα ευρωπαϊκά όργανα και δεν χρειαστήκαμε την συνεργασία των κρατών μελών στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά μόνο των ερευνητών δημοσιογράφων. Το θέμα της συνεργασίας με τα κράτη-μέλη είναι άλλη ιστορία, θα το συζητήσουμε σε άλλη αφορμή, για άλλες έρευνες, αλλά για μια ακόμη φορά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η ανάγκη εδώ είναι η έγκριση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τροπολογίας της Οδηγίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αυτό θα επιβάλλει σε όλα τα κράτη-μέλη και εδώ θα υπάρξουν αντιδράσεις ανάμεσά τους να δημοσιεύουν πληροφορίες οι οποίες θα μας επιτρέπουν να βρίσκουμε τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και ωφελούμενους από συγκεκριμένες ε, ε, χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες. Και έτσι όλα τα κρατημέλη θα αντιμετωπίζονται με ισότιμο τρόπο, χωρίς διαφοροποιήσεις. Θα ήθελα να συμμεριστώ την αισιοδοξία σας, λέει ο κύριος ε, Λάγγεν, αλλά παραμένουν κάποια ερωτήματα. Κύριε Ριοντέτ, νομίζω ότι αυτό σας αφορά ιδιαίτερα. Για τα έγγραφα του Παναμά. Θα πρέπει να προβλέψουμε <clears throat> ενέργειες συνεργασίες γιατί θα στείλουμε τα διάφορα πακέτα αναχώρα αυτή τη βδομάδα. Υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης, αλλά γενικά σε ό,τι αφορά τα θέματα λεύκανσης χρημάτων είναι πολύ καλή συνεργασία. Και πέρασα μια δύσκολη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω αυτού τα κράτη-μέλη έχουν κάθε θέληση και προθυμία να συνεργαστούν με τον ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ο Πάουλ Τάγκ και μετά δύο Catch the Eye της κυρίας Γκάμισ, Δεμάση και Λούκια και μετά πρέπει να κλείσουμε γιατί έχουμε το επόμενο πάνελ. Τάγκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τα μέλη του πάνελ για την παρουσία τους. Βλέπω ότι πολλά πράγματα είναι αλληλένδετα. Τα θέματα των περιπτώσεων φοροαποφυγής, έκπλησης χρημάτων κτλ. Ένα σημείο που ήθελα να τονίσω είναι το εξή. Όταν βλέπετε εσείς να υπάρχουν δίκτυα φοροαποφυγής, όταν κάνετε έρευνες από φοροαποφυγής που δεν είναι κατά παράνομη, αλλά που τις διακριβώνεται <clears throat> ούτως ή άλλως. Αναφέρεται κάτι τέτοιο στα κρατημέλη. Αυτό είναι ένα γενικό ερώτημα για το πάνελ. Ένα ειδικό ερώτημα για τον κύριο Ριοντέ. Βλέπουμε ότι κάποιες χώρες δεν παρέχουν πληροφορίες στο Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Κύπρος. ίσως δεν θέλετε να το απαντήσετε, αλλά γιατί δεν το κάνουν αυτό, τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες. Γιατί εσείς κάνετε κάποια προσπάθεια να διακριβώσετε γιατί αυτές οι χώρες δεν δίνουν τις ε, απαραίτητες πληροφορίες. Θα ήθελα να ξέρω την απάντησή σας. Και τι λένε όταν δεν δίνουν τις πληροφορίες αυτές. Ευχαριστώ. Ποιος θα ήθελε να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Από την Όλαφ και... Όχι, όχι. Δεν έχει τεθεί ερώτημα. Θέλετε να απαντήσετε κύριε Κάμπρη ή θέλετε να απαντήσετε γραπτός ή καθόλου. Την πρώτη σας ερώτηση. Ανάποδα πάει σε σχέση με το, τα στοιχεία τα οποία ερευνούν τα κράτη-μέλη. Εμείς δεν έχουμε ερευνητικές δραστηριότητες εμείς προσπαθούμε να συντονίσουμε τα στοιχεία τα οποία έρχονται από το ένα κράτος μέλος και το συνδυάζουμε με στοιχεία από το άλλο. Τι κάνετε σε περίπτωση που βλέπετε ίχνη ας πούμε φοροδιαφυγής. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω στατιστικές σε σχέση με αυτά. Συνήθως όμως η παρατήρησή σας ισχύει από την ανάποδη. συγγνώμη, ο κ. Σουριοντέ. για τα <clears throat> συστήματα αυτά φοροαποφυγής. Εμείς ερχόμαστε σε επαφή με τις ε, ομάδες υποστήριξης. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, κάποιες πάγιες πρακτικές που ακολουθούνται από, τρομο... από εγκληματικές οργανώσεις για φόρο το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σε σχέση με τη συνεργασία και με άλλα κράτη-μέλη. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει παροχή πληροφορίας, ίσα, ίσα δίδεται πληροφορίες, αλλά βέβαια μπορεί να βελτιωθεί η παροχή αυτή πληροφοριών. Εντάξει. Η Ρωμάνα Πανκ από το ΕΛΚ και μετά δύο Catch the Eye. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μας ενδιαφέρουν τα ίδια θέματα. Όλοι θέλουμε να ξέρουμε ποια κράτη-μέλη, ποιες χώρες είναι πιο συνεργάσιμες σε αυτή τη διαδικασία και ποιες είναι αυτές οι οποίες είναι πιο επιφυλακτικές σε σχέση με τη συνεργασία. Επειδή ετέθη αυτό το ερώτημα κάποιες φορές από τους ομιλητές, μου φαίνεται ότι δεν είσαστε έτοιμοι να μας δώσετε τα φώτα σας. Δεν θέλετε να δακτυλοδεικτήσετε και να μας πείτε ποιες χώρες δεν θέλουν να συνεργαστούν. Να αλλάξω τη μορφή αυτού του ερωτήματος. Θα το πω ως εξής. <clears throat> δεν είναι σωστό εμείς να μην επικροτούμε τη συμπεριφορά των χωρών αυτών που συνεργάζονται πλήρως. Πώς θα βελτιώσετε λοιπόν τη συνεργασία. Αν δεν θέλετε να μας πείτε ποιοι δεν συνεργάζονται, πείτε μας ποιοι συνεργάζονται. Ε, ο <laughs> κύριος ε, Κέσσερ δεν ξέρει ποιοι είναι καλοί μαθητές εδώ. Ε, απλή ερώτηση. Δεν συνεργαστήκατε με κανέναν, εμείς. Ε, μόνοι μας τα κάναμε. Ε, γιατί, όχι γιατί δεν μας αρέσει η συνεργασία. Δεν χρειαζόταν να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη. Όταν κάνουμε άλλες έρευνες για απάτες στον δημοσιονομικό τομέα, τον κοινοτικό, τότε πράγματι συνεργαζόμαστε με κράτη-μέλη. Αλλά αυτή είναι μια μακρά συζήτηση την οποία κάνουμε κυρίως με την ε, Επιτροπή Κοντ, ελέγχου προϋπολογισμών δηλαδή. Λοιπόν, για τα Panama Papers, ε, ό,τι χρειάστηκε να κάνουμε, τα κάναμε μόνοι μας χωρίς την παρέμβαση ουδενός. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και τώρα έχουμε τρεις ερωτήσεις του ενός λεπτού. Γιάννα Γκόμες. Ε, πρώτη, ένα λεπτό ερώτηση, δύο λεπτά απαντήσεις γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Να σας ρωτήσω το εξή. Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της, του καταλόγου των ε, εταιριών offshore με το σύνδεσμο με τις τρομοκρατικές οργανώσεις κτλ. και με τα κρατή-μέλη, γιατί δεν ε, νομίζω να μην υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος, ε, να μην υπάρχει τέτοια αναφορά. Και τι γίνεται όταν πηγαίνετε σε χώρες όπως η Γερμανία όπου υπάρχει απογοήτευση σε ό,τι αφορά τη νομική αρρωγή και τη νομική συνεργασία. Και μιλώ για συγκεκριμένε περιπτώσει όπου αφορά, για παράδειγμα, την πώληση υποβρυχίου στην Πορτογαλία, όπου ε, οι εμπλεκόμενοι καταδικάστηκαν στη Γερμανία, αλλά στην Πορτογαλία αυτοί που εμπλέκονταν δεν ε, εντοπίστηκαν ποτέ, γιατί υπήρξε συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και των υπετίων στην Πορτογαλία. Και αυτά υπογράφησε λοιπόν ε, επί ε, κυρίου Μπαρόσο. Και μία τέτοια αναφορά συμπεριλαμβάνεται και στα έγγραφα του Παναμά σε ό,τι αφορά μια εταιρεία με βάση τις Μπαχάμε και τον Παναμά. Μάλιστα. Θα δούμε ποιον θα ακούσουμε συγκεκριμένα και το έχει ξαναθέσει αυτό το ερώτημα σε ακρόαση η κυρία Γκόμε. Σιωπή που όμω επικρατεί στο πάνελ. Αν μου επιτρέπετε, δεν έχω να απαντήσω για την υπόθεση αυτή, την οποία την γνωρίζω πολύ καλά ασφαλώς, αλλά θα ήθελα επί της ευκαιρίας να πω το εξή. Αυτό που πάντα ερευνάμε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η, η έρευνα γίνεται με πολύ παροχημένο και παραδοσιακό, αν θέλετε, τρόπο πάντα από εθνικής οπτικής γωνίας, γιατί οι εθνικές αρχές είναι αυτές που πάντα ερευνούν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά το έγκλημα αυτό πολύ απλά δεν είναι εθνικό, είναι διαστοριακό. Σχεδόν όλες αυτές οι περιπτώσεις οι οποίες ερευνούνται δεν αφορούν έγκλημα το οποίο λαμβάνει χώρα σε μία μόνα χώρα. Γιατί η πραγματικότητα, η οικονομική πραγματικότητα και η εγκληματική πραγματικότητα είναι διασυνοριακή εκφύσεως. Αλλά εμείς εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε τις τακτικές του 19ου αιώνα. Κατακαιρματισμένη η έρευνα. Αυτό λοιπόν είναι ένα σαφές παράδειγμα του πόσο παροχημένη είναι η μέθοδος έρευνάς μας και του πόσο χρειάζεται κάτι επιγόντως μια ευρωπαϊκή διάσταση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δρά ως ενιαίος χώρος. Όσο το πετυχαίνουμε αυτό, πάντα θα ψάχνουμε να βρούμε τον καλό και τον κακό το μαθητή και ουσιαστικά θα να για μια πιο καλή συνεργασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φάβιο Ντιμάζη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση προς τον κύριο Ριοντέ. Δουλεύει το μικρόφωνο μου. Μία ερώτηση προς τον κύριο Ριοντέ από τη Γερεπόλ. Στις απαντήσεις σας είπατε ότι είχατε κάποιες χιλιάδες hits ε, σε ό,τι αφορά τη βάση δεδομένων για τα Panama Papers και υπάρχουν κάποια focal points, κάποια σημεία σε Το Hydra, το Ισλαμικό τρομοκρατικό δίκτυο και είπατε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν τα πιο πολλά hits ή πιο πολλές τέτοιες ε, ευρέσεις. Ε. Σε ό,τι αφορά τον παγκόσμιο Ισλαμικό τρομοκρατικό κύκλο, ποια χώρα είχε τα πιο πολλά hit και επειδή είμαι Γερμανός ε, βουλευτής μας ενημέρωσε η σχετική γερμανική αρχή ή το Σώμα Οικονομικού Κλίματος μας ενημέρωσε λοιπόν ότι ένα πρόβλημα είναι που υπάρχει έλλειψη ε, για μια βάση δεδομένων για τα κτηματολόγια. Ο κύριος Ριοντέ, δύο λεπτά για τις απαντήσεις. σχετικά με τις τρομοκρατικές δραστηριότητες. Είχαμε 160 hit σχετικά με τις χώρες που παρέχουν πληροφορίες στη Europol. Εμείς προστατεύουμε τα δεδομένα φυσικά και προστατεύουμε και τα δεδομένα και τα συμφέροντα των κρατών μελών, ως εκ τούτου δεν απαντώ στην ερώτησή σας data protection. Uh, uh, Όχι μόνο μονομένων προσώπων, όπως γνωρίζετε στη Europol τα στοιχεία προστατεύονται σύμφωνα με την βούληση αυτών που μας τα παρέχουν. Και γι' αυτό ακριβώς φτιάχνουμε αυτά τα πακέτα και τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία επιλέγουν τι είναι δημοσιεύσιμο και τι όχι. Για τον κύριο Ντεμάζη. Ζητώ την κατανόησή σας. Εγώ ως εκπρόσωπος ενός οργάνου της Ένωσης δεν μπορώ να κάνω κριτική ή σχόλια στο τι αποφασίζεται στα κράτη-μέλη. Το θέμα είναι ότι η Eurojust θέλει μέσω του συντονισμού να ξεπεράσει τις διαφορές που υπάρχουν στα εθνικά συστήματα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, εμείς εργαζόμαστε. Το θέμα δεν είναι να επιλέγουμε τις ε, καλές ε, μορφές ενημέρωσης, το θέμα είναι να εκμεταλλευόμαστε μέσω του συντονισμού όλες τις μορφές ε, ενημέρωσης. Αυτό είναι το πρέπον και αυτό κάνουμε. Χωρίς, χωρίς μικρόφωνο. Κύριος Λούκε και έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας νομίζω ήδη. Ένα σύντομο ερώτημα. Εμείς είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών και μας αρνείτε να μας δώσετε στοιχεία για ένα ερώτημα το οποίο είναι απόλυτα θεμητό σε σχέση με τη σύνδεση με τρομοκρατία. Αυτό είναι απαράδεκτο για μένα. Και το ερώτημα στο οποίο ήδη είχε θέσει ο κύριος Λάγκεν. Θα ήθελα να θέσω για τις χώρες. Θα ήθελα να θέσω ερωτήματα για την Αυστρία και το Λουξεμβούργο που έχουν μια εξαίρεση από την οδηγία για τον ευρωπαϊκό, για την φορολογία των αποταμιεύσεων. Είναι αλήθεια ότι το Λουξεμβούργο και η Αυστρία συνεργάζονται στον ίδιο βαθμό όπως οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι. Ευχαριστώ, παρακαλώ. Ποιος θεωρεί ότι μπορεί να απαντήσει στο θέμα αυτό. Μα θα ακούσουμε και τους εκπροσώπους των χωρών αυτών στη συνέχεια. Όχι. Δεν μπορείτε να, να λάβετε θέση κύριε Κάμπρη. Σας είπα κύριε Λούκε ότι για τα έγγραφα του Παναμά έχει λάβει χώρα η μεγαλύτερη διαδικασία συντονισμού που έχουμε γνωρίσει. Υπάρχει λοιπόν η θέληση των κρατών μελών να συνεργαστούν και σταματώ εδώ. Κύριε Ζήοντε, δεν υπάρχει κάποια απάντηση από την Ιεροπόλ. Κύριο Κέσλε. Δεν είναι ότι δεν θέλω να πω, είναι το ότι είπα ότι εγώ δεν συνεργάστηκα για το ε, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με τα κράτη-μέλη. Είναι εκτός αρμοδιότητάς μου. Ως εκ τούτου εγώ δεν ασχολήθηκα με αυτό μαζί με τα κράτη-μέλη. Εγώ έχω συνεργαστεί με το Λουξεμβούργο για άλλου είδους απάτες και άλλου είδους ε, ποινικέ ε, διαδικασίες και οι χώρες αυτές συνεργάζονται όπως και όλες, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα, για το ξέπλυμα, για τη φοροδιαφυγή, αυτά είναι εκτός αρμοδιοτήτων μου. Με καμία χώρα δεν συνεργάζομαι γύρω από αυτό το θέμα. Ζητώ συγγνώμη. Οι συνάδελφοί μου είναι σε διαφορετική κατάσταση από μένα. Πρέπει να βρούμε ένα άλλο τρόπο για να απαντηθεί το ερώτημά σας, λέει ο κύριο Λάγκελ. Ευχαριστώ και τα τρία μέλη του πάνελ που μας ε, διαφώτισαν. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο ακούσαμε. Είχαμε, διαπιστώσαμε ότι γενικά είναι καλή η συνεργασία για τα έγγραφα του Παναμά και θα προσπαθήσουμε και στη συνέχεια να απαντήσουμε τα ερωτήματα τα οποία παρέμειναν εκκρεμεί. Ευχαριστώ τον κύριο Μάιερ Κάμπρι, τον κύριο Ριοντέ και τον κύριο Κέσλερ. Δύο λεπτά διάλειμμα για, για να έλθει το επόμενο πάνελ. Ah, voilà, je vais me déconnecter. Je vous laisse. Merci. Désolé. Hein.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 Κυρίε και κύριοι, να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε με το δεύτερο τμήμα. Πέντε η ώρα αντί για πέντε παρά τετάρτο, όπω προβλεπόταν. Αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια. Να είμαστε πιο σύντομοι στι ερωταπαντήσει. Και θα ήθελα να ορίσω στο πάνελ τον κύριο Φίλιπ Τεκώστερ, πρόεδρο της ε, Βελγικής ε, Υπηρεσίας Καταπολέμησης Οικονομικού Κλίματος και τον κύριο Μισελ Κλέζ. Πού πήγε? Εδώ τον είχα. Μάλιστα. Εισαγγελέα από το Βέλγιο, Νόρμπερτ Ναουλίν, ο οποίος είναι επικεφαλής της ε, Υπηρεσίας Ειδικών Ερευνών ΕΟΚΣ, ομάδα ερευνών οργανωσμένου εγκλήματος από την Βόρεια Ευδανία Βεσφαλία. Ο οποίος ε, έλαβε υπόψη της ε, τα του Παναμά. Και πρέπει να σας πούμε ότι στην βιντεοδιάσκεψη ε, είναι λίγο, έχουμε μια έλλειψη φωτεινότητας αλλά βλέπουμε τον κύριο Πάτρικ Μοντανιέ, ο οποίο είναι μέλος του σώματο των γαλλικών εποπτών. Σα καλωσορίζουμε λοιπόν και τους τέσσερι. Έφυγε ο κύριος ε, από το Βέλγιο, ο γενικό Εισαγγελέα. Εν πάση περιπτώσει, θα ξαναμπεί μέσα, ελπίζω. Ξεκινούμε. Σα καλωσορίζω Χωρί ε, εισαγωγικά σχόλια, γιατί δεν έχουμε και χρόνο, έχουμε καθυστερήσει και θα το εκτιμούσα ιδιαίτερω αν μπορούσατε να περιοριστείτε στα 8 λεπτά αντί για 10 λεπτά, προκειμένου να ακούσουμε και τις ερωτήσεις μετά. Καλώς ήρθατε και εσείς κύριε Κλέζε. Και θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα-πρώτα στον πρόεδρο της Βελγική Υπηρεσίας Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος τον κύριο Φίλιπ Τεκόστερ, για το πώς αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό σε εθνικό επίπεδο. Ποιες είναι οι παρουσιάσεις σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Μπορώ να μιλήσω σε τρεις γλώσσες και γι' αυτό θα μιλήσω γαλλικά που δεν άκουσα και πολύ σήμερα το απόγευμα. Προετοίμασα ένα έγγραφο και θα μείνω στα οκτώ λεπτά, Πρόεδρε. Είμαι υπεύθυνο ε, για ένα κέντρο Βελγικό Συλλογή Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πληροφοριών. Να σας δώσω μια μικρή περίληψη αυτού το οποίο κάνουμε και για να ξεφύγω από το κείμενό μου και νομίζω ότι είχα κάποια στοιχεία να συνεισφέρω σε σχέση με τα Panama Papers. Λοιπόν, το κέντρο αυτό δημιουργήθηκε το 1993. Από το 1995 και μετά, έτσι, ε, καταπολεμούμε το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διότι δεν είναι καινούριο πράγμα για μας και οι φορολογικές απάτες μετά για 7-8 χρόνια ε, κλεπτύναμε αν θέλετε αυτήν την εξωτική κατά τα άλλα έννοια για να περιοριστούμε στις σοβαρές οργανωμένες εφοριακές απάτες. Νομίζω ότι κατανοείται ότι οι απλές φορολογικές απάτες δεν ανήκουν πλέον στις αρμοδιότητές μας. Λοιπόν, τι κάνει αυτό το κέντρο συλλογής πληροφοριών το Βελγικό υποδέχεται, λαμβάνει κάποιες δηλώσεις υπόπτων περιπτώσεων είτε Βέλγων είτε Βελγικών εταιριών είτε εταίρων τους στον υπόλοιπο κόσμο και προχωρά σε κάποιες αναλύσεις αυτών των αναλύσεων ή δηλώσεων υπόπτων συναλλαγών. Έχουμε τη δυνατότητα εμείς να συμβουλευτούμε όλες τις υπηρεσίες του κράτους δηλαδή τις δικαστικές αρχές, τις αστυνομικές αρχές, την κατασκοπία, τις φορολογικές αρχές. Έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε την άποψη της ΟΛΑΦ όταν κάτι γίνεται εις βάρος του προϋπολογισμού του κοινοτικού. Έχουμε λοιπόν μια διευρυμένη αρμοδιότητα και εξουσία αν θέλετε, όταν μια συναλλαγή μας φαίνεται ύποπτη Έχουμε την ευθύνη και το καθήκον να μεταφέρουμε στις δικαστικές αρχές τον φάκελο και ταυτόχρονα στο Βέλγιο έχουμε την δυνατότητα να, να δεσμεύσουμε διοικητικά ε, λογαριασμούς και συναλλαγές για πέντε εργάσιμες ημέρες. Ένα παράδειγμα. Αν την προηγούμενη Δευτέρα ήθελα να δεσμεύσω τους λογαριασμούς ενός προσώπου, μπορούσα να το κάνω για πέντε μέρες. Αυτή λοιπόν η προσωρινή δέσμευση σταματάει αύριο γιατί την προηγούμενη Παρασκευή δεν ήταν καθημερινή ημέρα και μετράμε μόνο τις εργάσιμες. Ε, Ένα από τα θέματα τα οποία τέθηκαν είναι και ε, το ξέπλυμα και η φορολογική απάτη. Το ξέπλυμα πάρα πολλών προσόδων από οικονομικές δραστηριότητες. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε κάποιες βασικές παραβάσεις οι οποίες προκαλούν κάποια κέρδη και τα κέρδη αυτά είναι αυτά τα οποία την χάνουν ξεπλήματος. Μπορεί να υπάρχουν φορολογικές απάδες, το προϊόν αυτής της φορολογικής απάτης μπορεί να κατευθυνθεί σε ένα λογαριασμό σε οποιαδήποτε χώρα ή να μετατραπεί σε αγαθό, κινητό ή ακίνητο Έχουμε την δυνατότητα λοιπόν καταπολεμώντας το ξέπλυμα και να δεσμεύσουμε λογαριασμούς και ε, κατά περίπτωση να μεταφέρουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα οδηγήσουν σε ε, τέτοια δέσμευση. Γιατί να καταπολεμούμε λοιπόν το ξέπλυμα, όπως, είμαι και, όπως σας είπα είμαι και εισαγγελέα, έχω το βαθμό εισαγγελέα. Έχω την πεποίθηση λοιπόν εδώ και πολύ καιρό ότι στον τομέα των χρηματοπιστωτικών πρέπει να αναπτύξουμε μια κάποια στρατηγική. Εγώ σαν μέλος της υπηρεσίας μου θα μπορώ να προχωρήσω στη δίωξη του ξεπλήματος προσόδου από οποιοδήποτε εγκληματική δραστηριότητα. Αλλά υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι, δικαστές, εισαγγελείς, αστυνομικοί, οι οποίοι αναζητούν τα στοιχεία των βασικών παραβάσεων, δηλαδή οικονομική εγκληματικότητα, οργανωμένο έγκλημα, σωματεμπορία, πορνεία τι είναι από όλα αυτά το πιο σημαντικό, η καταπολέμηση του ξεπλήματος ή οι αρχικές παραβάσεις. Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτή τη στιγμή συλλάβουμε τους ε, υπόπτους, αυτό δεν το κάνουμε δυστυχώς πάντα γιατί μπορεί να έχει παρέλθει, να έχει επέλθει παραγραφή. Ανάλογα με την δραστηριότητα αλλά το ξέπλυμα μπορεί εκ των υστέρων να χρησιμοποιηθεί, είναι μια ασφάλεια την οποία έχουμε στον χρόνο, μια ρήτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να επιβάλλουμε κυρώσεις όχι λόγω μιας παράβασης ποινική, αλλά λόγω, αν θέλετε, της δραστηριότητάς του της οικονομικής εκ των υστέρων. Να επανέλθω τώρα σε αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει, στα Panama Papers και τη φορολογική απάτη. Απλή ή σοβαρή, οργανωμένη ή όχι. Είχαμε την δυνατότητα να συνεργαστούμε με τις διοικητικές υπηρεσίες, τις φορολογικές στο Βέλγιο. Είδαμε τους ελέγχους σε επίπεδο ΦΠΑ. Τους ζητάμε πληροφορίες, τους ζητάμε στοιχεία και μας δίνουν στοιχεία που τροφοδοτούν τις δικές μας αναλύσεις. Δεν έχουμε λοιπόν φόβους όταν ασχολούμεθα με θέματα ξεπλήματος που προέρχονται από φορολογικές παραβάσεις. Αλλά όταν μιλάμε για φορολογικές απάτες πρέπει να κάνουμε διαφορετικές εδώ διακρίσεις. Πρώτον, η απάτη στο ΦΠΑ είναι απλή και ανακαλύπτεται αμέσως. Και έρχομαι σε κάτι που σας ενδιαφέρει. Οι λογαριασμοί offshore στον Παναμά, σαν παράδειγμα, το ότι έχει κανείς κάποιον στο εξωτερικό, αυτό, αυτό δεν είναι παράβαση. Αλλά το ότι δεν το δηλώνει όταν καταθέτει, θα έλεγα, μια φορολογική δήλωση, γίνεται παράβαση. Ο συνάδελφός μου σαν παράδειγμα που τον γνωρίζω καλά ανοίγει ένα λογαριασμό στις Μπαχάμες. Αυτό δεν είναι παράνομο. Αν τον επόμενο χρόνο όμως όταν καταθέτει τη φορολογική του δήλωση δεν δηλώνει τον λογαριασμό αυτό τότε είναι. Και εκεί ξεκινάει μια δικασία. Μέχρι σήμερα λοιπόν για 5-6 μήνες ε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ε, περιμένω να κάνει ε, μια στραβή σε εισαγωγικά ο παρακαθήμενος για να μπορέσω και εγώ να δράσω. Ξεφεύγω από το εθνικό κομμάτι, <clears throat> μιλάμε για τις αποκοινές προσπάθειες που γίνονται από την Eurojust και από την ε, Europol. Ξέρω για τις μορφές ε, συνεργασία. Υπάρχει συνεργασία με 7 υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών το Βέλγιο είναι καλός μαθητής νομίζω συνεργάζεται με την Ευρωπόλ. Υπάρχουν άλλες χώρες, όχι που δεν συνεργάζονται, αλλά που έχουν κάποιους δισταγμού. Πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, υπάρχει ένα πλαίσιο εδώ, υπάρχει ένα σώμα, το, η ομάδα EGMO, η ομάδα ΕΓΜΟ αντιπροσωπεύει 180 υπηρεσίες συλλογής οικονομικών στοιχείων. Γιατί ΕΓΜΟ, γιατί η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε από τους Βέλγους και τους Αμερικανούς το 1995 στο Παλέντε ΕΓΜΟ εδώ στις Βρυξέλλες, εξ αυτού το όνομα. Όλες λοιπόν αυτές οι υπηρεσίες συλλογής οικονομικών πληροφοριών συναντώνται τρεις-τέσσερις φορές το χρόνο για να συζητήσουν τα θέματα αυτά και φυσικά συμμετέχει και ο Παναμάς. Ας επανέλθουμε τώρα κύριε Πρόεδρε στο θέμα του Παναμά. Πήρα ονόματα, μου έστειλαν ονόματα οι φορολογικές αρχές 240 και ο οργανισμός μου μέχρι σήμερα έχει ξεκινήσει 97 φακέλους. Τι βλέπω για αυτούς τους φακέλους, τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω γιατί ζήτησα από τον Παναμά να μου δώσει συμπληρωματικές πληροφορίες, ε, δεν απελπίζομαι, περιμένω, έρχονται Χριστούγεννα, μπορεί και οι Παναμέζοι να μου κάνουν ένα δώρο. Πάντως, κάτι κάνουμε με τα μέσα τα περιορισμένα που έχουμε. Πέντε δευτερόλεπτα ακόμα για να μιλήσω για συνεργασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε συνέργειες και μπορεί ίσως να σας σοκάρω γιατί γίνεται αυτό συχνά θα ακούσαμε να μιλάμε για την ε, Eurojust, την Europol, γιατί να μην συζητήσουμε την δημιουργία ε, μιας ε, ειδική υπηρεσίας καταστολής της φορολογικής απάτης ευρωπαϊκής. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος <clears throat> Μονταγέ, ο οποίος είναι συνδεδεμένος μαζί μας με το κ. Μοτανιέ, ο οποίος είναι μέλος του Γαλλικού ε, Σώματος ε, Εποπτών, θα συνδεθεί μαζί μας με βίντεο και θα λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Νομίζω ότι είναι κάπως σκοτεινή η εικόνα από τη δική σας πλευρά. Από τη δική μου πλευρά είναι μια χαρά βέβαια. Πάρα πολύ σύντομα θέλω να σας υπενθυμίσω τι είναι η Γαλλική Αρχή ελεγκτών. Δημιουργήθηκε το 2010 με την συγχώνευση των ε, εποπτικών φορέων των τραπεζών και άλλων φορέων. Έχουμε τρεις κύριες αποστολές. Τον προληπτικό έλεγχο, δηλαδή το να εξασφαλίσουμε ότι λειτουργούν σωστά οι κανόνες πρόληψης, επίσης τον αγώνα κατά της ε, λεύκανσης χρημάτων και κατά της χρήσης των κονδυλίων αυτών από την τρομοκρατία, που θα επανέλθω στο θέμα αυτό, και τρίτον, ο στόχος μας είναι να ελέγξουμε τις εμπορικές ε, ε, δραστηριότητες των <clears throat> τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών. Υπάρχει μια αρχή χρηματαγορών που ελέγχει την, ε, τις συναλλαγές στα χρηματιστήρια και τις πωλήσει αξιογράφων από τις τράπεζες ανεξάρτητα από τη μορφή των πολιτών και αγοραστών. Εμείς λοιπόν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα των εγγράφων του Παναμά. Εκεί εμπλέκεται η δική μας ευθύνη για τη λεύκανση χρημάτων και καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είναι δύο σημαντικοί άξονες για μας. Είναι σαφές ότι η αρχή ελέγχου έχει ένα ρόλο για να εξασφαλίσει ότι οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και η ενδιάμεσή τους σέβονται απόλυτα την νομοθεσία. Δεν είμαστε βέβαια μια αρχή για τη συλλογή πληροφοριών στη Γαλλία, όπως ε, στην περίπτωση του προηγούμενου μιλητή για το Βέλιο. Είμαστε ο φορέας ο οποίος ασχολείται με τον ε, συγκεκριμένο τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα και την εφαρμογή της νομοθεσίας στα θέματα αυτά. Κάνουμε ορισμένους ελέγχους είτε εξ αποστάσεως είτε επιτόπου. Ο έλεγχος εξ αποστάσεως είναι πιο μόνιμος, μας επιτρέπει να εξασφαλίσουμε ότι <clears throat> τα έγγραφα σε σχέση με τη δημιουργία κάποιων διαδικασιών στις τράπεζες αυτές έρχονται σε εμά. Έχουμε επίσης και δειγματοληπτικές έρευνες κάθε χρόνο για να ελέγξουμε ορισμένε ε, καταστάσεις. Ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξουμε όμως είναι να κάνουμε επιτόπιες έρευνες ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι διαδικασίες όπως μας περιγράφονται από τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες λειτουργούν πράγματι και επιτρέπουν στους φορείς αυτούς να φέρουν σε πέρα στο καθήκον της διαπίστωσης της ταυτότητας των ε, πελατών τους και επίσης τη δήλωση υποψιών όταν είναι απαραίτητο ενώπιον της αρμόδιας αρχής στη Γαλλία. Για τα έγγραφα του Παναμά <clears throat> που ζητήσατε να έχετε περισσότερες λεπτομέρειες από εμά και εμείς έχουμε διατυπώσει ένα πιο πλήρες έγγραφο, έχουμε ξεκινήσει μια σειρά από έρευνες ήδη από τον Απρίλιο του 2016 έναντι όλων των τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό ή διαχειρίζονται ιδιωτικά κεφάλαια για να ξέρουμε αν από την πλευρά των πελατών τους υπήρξαν συνδέσεις με τις εταιρείες αυτές στον Παραμά που δημιουργούν εταιρείε offshore και επίσης Αυτές είναι πληροφορίες που προσπαθούμε ακόμα να αξιολογήσουμε πλήρως. Υπήρξαν πάνω από 100 email που έχουμε στείλει για να πάρουμε πληροφορίες και επίσης προσπαθούμε <clears throat> να δούμε τι πρέπει να κάνουμε εναντί κάποιων φορέων που έχουν αναφέρει ότι έχουν κάποιες διασυνδέσεις με τα έγγραφα του Παραμά ή χρειάζονται περαιτέρω ε, έρευνα. Θα υπάρξει λοιπόν μια έκθεση για τα θέματα αυτά που θα γίνουν ε, <clears throat> από τις αρμόδιους φορείς ή αλλιώς εμείς θα προβούμε σε μια σειρά από ελέγχους σε σχέση με τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε ε, διεθνές επίπεδο για να δούμε αν υπάρχει πράγματι λόγος περαιτέρω έρευνας μετά από τις πρώτες μας επαφές με τις ε, τραπεζικές αρχές. Σε ό,τι αφορά το την φοροδιαφυγή δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο το θέμα της λεύκανσης χρημάτων και ε, τρομοκρατίας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε όμως ότι τα τραπεζικά και ασφαλιστικά ιδρύματα θα περιλάβουν και τη φοροδιαφυγή μεταξύ των αδικημάτων που μπορούν να δώσουν λαβή σε λεύκανση χρημάτων. Στη Γαλλία το να τεθεί η φοροδιαφυγή στα υποκείμενα αδικήματα που μπορούν να προκαλέσουν το ξέπλυμα χρημάτων ήταν πολύ σημαντικό, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί ο αγώνας κατά της φορολογικής φοροδιαφυγής μπορεί να ε, βοηθήσει την αντιμετώπιση τη λεύκανση χρημάτων, παρά το γεγονό ότι αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχει αντιμετωπιστεί πλήρω από όλε τι χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν και μια σειρά εργαλείων για του ελέγχου μα. Είναι πολύπλοκη αυτή η διαδικασία, αλλά ο στόχο μα θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε ένα αποτελεσματικό έλεγχο των πολυεθνικών ομήλων. Εμείς είμαστε αρμόδιοι για να εξασφαλίσουμε ότι οι φορείς αυτοί που βρίσκονται στην Γαλλία, είτε παροχή υπηρεσιών, οι τράπεζες και ασφάλειες εγκατεστημένες στη Γαλλία ή με μορφή θηγατρικών, σέβονται πλήρως τη γαλλική νομοθεσία. Όταν πρόκειται για υποκαταστήματα και θηγατρικές γαλλικών τραπεζών πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάλι θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια γενική σωστή αντιμετώπιση από τους ομίλους αυτούς που σέβονται και πάλι την νομοθεσία και θέλουμε <clears throat> πάντα να τους, πάντα τους ζητούμε να μας δηλώσουν σε ποιες χώρες υπάρχει νομοθεσία η οποία μπορεί να αποτελέσει πρόσκομα στην τήρηση των υποχρεώσεών τους βάσει της γαλλικής νομοθεσίας. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να γνωρίζουμε να γνωρίζουν οι μητρικές εταιρείε τι ακριβώς συμβαίνει με τις θηγατρικές. Σε ορισμένε περιπτώσει η ιστορία δείχνει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και πολλές φορές έρχεται σε σύγκρουση το τραπεζικό ε, απόρριτο στην παράδοση, στην παροχή πληροφοριών ακόμα και στις μετρικές εταιρείε. Προσπαθούμε επίσης να συνάψουμε συμφωνίες με ξένες, ε, ε, με δικαστικές αρχές τρίτων χωρών για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Τονίζουμε ότι η πάταξη της λεύκασης χρημάτων έχει να κάνει με τη χώρα που λαμβάνει η χώρα το αδίκημα. Εμάς μας ενδιαφέρει η διάδεση μεταξύ της θηγατρικής και της μιτζικής εταιρεία στη, Γάλα, στη Γαλλία και την ανάγκη να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίε στον επόπτη στη Γαλλία. Αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε θηγατρικές άλλων εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι απλώς στην περίπτωση που υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα να επιβάλλουμε κυρώσεις στη μητρική εταιρεία για το γεγονός ότι δεν έχει τον έλεγχο πάνω στις θηγατρικές της εταιρείε και τα υποκαταστήματα και βέβαια δεν μπορούμε να τις κολλάσουμε για το γεγονός ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο δίωξης στις χώρες αυτές. Έχουμε επίσης την ικανότητα να ενισχύσουμε τις ε, ε, διατάξεις σε σχέση με την ε, λεύκανση των χρημάτων, διότι έχουμε διτό χαρακτήρα ως επόπτες και ως αρμόδιοι για τα θέματα λεύκανσης χρημάτων. Ο τρόπος με τον οποίο οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες ο τρόπος με τον οποίο διαθρώνουν τους ελέγχους τους είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αν γίνεται αυτό με τρόπο σύμμορφο με αυτά που είναι απαραίτητα για την πάταξη τέτοιων δραστηριοτήτων όπως η λεύκαση χρημάτων δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποχωριστεί από τις υπόλοιπε δραστηριότητες των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι τμήμα της καθημερινής εμπορικής δραστηριότητά του με του, των πελατών του, Όλα ξεκινούν με τον εντοπισμό το, της ταυτότητας των πελατών τους και των ποσών που μπορούν να διακινηθούν από την τραπεζική ή ασφαλιστική λειτουργία για τους πελάτες τους. Έχουμε λοιπόν κάποιες ε, συνδέσεις με το κέντρο χρηματοπιστωτικών πληροφοριών στη Γαλλία. Πολλές φορές μας παραπέμπει περιπτώσεις οι οποίες φαίνεται ότι ε, εμπίπτουν σε υποψία έλλειψης ελέγχου για τις συναλλαγές Είμαστε σε επαφή επίση για τα φορολογικά θέματα με τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οικονομικών στη Γαλλία, στην οποία μετα... <clears throat> μεταφέρουμε πάντα, διαβιβάσουμε τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων μας. Βέβαια, δεν ασχολιόμαστε με ειδικέ περιπτώσει απάτης στι δεκάδε χιλιάδε συναλλαγών που γίνεται κάθε φορά, αλλά κάνουμε ελέγχου για να δούμε αν λειτουργεί ο μηχανισμό λαμβάνουμε υπόψη στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποια υποψία και αν αυτή η υποψία έχει να κάνει με ένα κίνδυνο φορολογικής απάτης, το παραπέμπουμε στην ε, αρχή των, την ε, Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Θεμάτων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μοντανιά. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση των πρακτικών που ακολουθούνται στη Γαλλία και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο θα δώσω το λόγο κατευθείαν προς τον κύριο Μισελ Κλέζ στον εισαγγελέα από το Βέλγιο για να μας ε, παρουσιάσει τις αρμοδιότητές του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν είμαι εισαγγελέα, είμαι δικαστής ερευνητής. Και γι' αυτό θα σας μιλήσω ακριβώς ανεξαρτήτως από τις απόψεις της εισαγγελία. Η εμπειρία μου μετά από τόσα χρόνια μου επιτρέπει να σας πω καταρχάς ότι μαθαίνοντας ε, για τα Panama Papers προσεκλήθηνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της χώρας μου και τους είπα ότι εγώ δεν εκπλήσωμαι, εσείς γιατί εκπλήσεστε. Εδώ και πολύ καιρό όσοι καταπολεμούν την ε, εγκληματικότητα σε οικονομικό επίπεδο γνωρίζουν το φαινόμενο αυτό και Μάθαμε για τα Panama Papers, αλλά του χρόνου θα έχουμε τα Tortola Papers, μετά τα Cayman Papers και Μπαχάμες και δεκαετίες μας περιμένουν με τέτοιου είδους ετήσια σκάνδαλα. Το θέμα είναι το φαινόμενο αυτό να σταματήσει να λειτουργεί και αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί αν στο Βέλγιο, γιατί γι' αυτό μιλάω, ε, δεν μάθαμε και πάρα πολλά πράγματα για τις δραστηριότητες αυτών των ανθρώπων στον Παναμά, αλλά παρόλα αυτά το φαινόμενο μας επιτρέπει να έχουμε κάποιες επιτροπές στη διάθεσή μας και ίσως στο μέλλον κάποιες αντιδράσεις που να έχουν νόημα και έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Ε, σε σχέση με αυτά το οποία είπε ο Φιλίπ Ντεκοστέρ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο φορολογικό και το να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, αν θέλετε, ε, τα Panama Papers θα πρέπει να τα θεωρούμε σαν εγκληματική οικονομική δραστηριότητα και όχι σαν φοροδιαφυγή. Έχετε τέσσερις τύπους παρατυπιών στον τομέα της ε, οικονομικής δραστηριότητας. Καταρχάς είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πολύ νομικές, ε, πολύ ένομες θα έλεγα, παρουσίες φυσικές έχετε ας πούμε κάποιο πρόβλημα υδραυλικό, φωνάζετε κάποιον να σας το φτιάξει, δεν κόβει απόδειξη. Ε, εντάξει, είναι μια μικρή απάτη. Η δεύτερη απάτη είναι να φτιάξετε μια μικρή πισίνα και τα χρέη να, να χρεωθεί η επιχείρησή σας και όχι εσείς, παρότι είναι προσωπική. Το τρίτο στάδιο είναι η διαφθορά. Έχουμε και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα λιγότερο από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. Ίσως είναι ενδημικό φαινόμενο το οποίο εμποδίζει τις δημοκρατίες να επιβιώσουν. Αυτό το φαινόμενο της διαφθοράς υπάρχει και αυτή είναι ποινικά κολάσιμη δραστηριότητα ανθρώπων που έχουν μια νόμιμη παρουσία στην κοινωνία. Και η επόμενη φάση είναι οι λεγόμενες μεγάλες παραβάσεις του κοινού δικαίου. Εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε για την οικονομική ε, δραστηριότητα η οποία όμως θα έλεγα πολλές φορές γίνεται ιονή. Από ό,τι λένε ε, ε, αυτή τη στιγμή ξεπλένονται 250 εκατομμύρια το χρόνο στην Ευρώπη με βάση κάποιες μη υπάρχουσες ουσιαστικά συναλλαγές. Γίνονται απάτες online στο διαδίκτυο, ε, επίσης κάποιες εταιρείες ε, ε, λειτουργούν σαν εγκληματικές συμμορίες και βγάζουν χρήματα από τις φορολογικές υπηρεσίες των κρατών μελών ε, και νομίζω ότι πάρα πολλά χρήματα που χάσαμε εδώ στο Βέλγιο πήγαν στο Ντουμπάι, κάτι το οποίο δεν θα μας κάνει να τα δούμε ξανά. Ε, και επίσης υπάρχουν ε, και κέρδη από, από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, από τα παραποιημένα προϊόντα, 35 εκατομμύρια το χρόνο, από το λαθρεμπόριο όπλων, από τη σώματεμπορία. Όλες αυτές οι σοβαρές μορφές ε, οικονομικής εγκληματικότητας παράγουν βρώμικο χρήμα το οποίο ανακυκλώνεται. Ένας τρίτος τύπος είναι η τρομοκρατία φυσικά έχει κάποια ειδικά ε, χαρακτηριστικά γιατί η οικονομική παράβαση γίνεται εκ των προτέρων και μετά ακολουθεί η τρομοκρατική ενέργεια. αλλά προφανές είναι ότι δεν υπάρχουν μόνο τα θέματα του, του, των ενεργειών των τρομοκρατικών, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα άλλου είδους όπως η ριζοσπαστικοποίηση κτλ. Και από την άλλη έχουμε και τους ενδιαμέσους, αυτούς οι οποίοι διαμεσολαβούν. Πολλές φορές είναι τράπεζες, είναι οικονομικοί σύμβουλοι, φορολογικοί σύμβουλοι, ορκωτοί λογιστές, δικηγόροι, για να είναι κανείς αποτελεσματικός για την καταπολέμηση φαινομένων όπως τα Panama Papers, όλοι αυτοί είναι αυτοί τους οποίους θα πρέπει να εντοπίσουμε. Θα μιλήσω σαν Βέλγος, θα μπορούσα επί μία ώρα να σας πω ότι η πολιτική μου στον τομέα αυτό της χώρας μου δεν είναι καθόλου καλή. Θα προσπαθήσω όμως να είμαι θετικός και να πω ότι υπάρχει μια αριθμιστική δυνατότητα παρέμβασης που έχουμε στον τομέα του ξεπλήματος, σαν παράδειγμα. Μετά από τον εξαιρετικό νόμο εντοπισμού που, στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Ντεκοστέρ, ο οποίος επιτρέπει να βρίσκουμε τις ύποπτες συναλλαγές. Έχουμε επίσης και τον, το άρθρο 105 του ποινικού κώδικα που συστήνω σε όλες τις χώρες ε, όπου θεωρείται κύρια η οικονομική ποινικά κολάσιμη δραστηριότητα το ξέπλυμα και όχι δευτερεύουσα. Η κατάσχεση η δέσμευση και μετά η κατάσχευση των προϊόντων μιας εγκληματικής δραστηριότητας γίνεται κατά αναλογία. Ε, ε, δεν ε, ίσως βρίσκουμε απευθείας το ίδιο το προϊόν της συναλλαγής, αλλά θα έλεγα τις συνέπειες του προϊόντος αυτού. Νομίζω λοιπόν ότι έτσι μπορούμε αυτού του είδους τις νομοθετικές δραστηριότητες και πρέπει να τις επιβάλλουμε παντού. Έχω λίγα λεπτά ακόμα, θα ήθελα να πω σαν εκπρόσωπος ευρωπαϊκής χώρας ότι πολλά μένει να γίνουν ακόμα και τέρα. Τα είπε ο κύριος Ντεκοστέρ. Το 2011 το Φεβρουάριο είχα πάρει μέρος στις συναντήσεις που κάναμε ε, στην Χάγη στα πλαίσια του Eurofisk. Είναι ένα κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι θα έλεγα χρήσιμο και αποτελεσματικό ε, για το ε, πανηγύρι αν θέλετε της ΦΠΑ, της απάτες του ΦΠΑ. Οι φάσεις τις οποίες πρέπει να περάσουμε τα στάδια είναι από τη μία να εντοπίσουμε το modus βοπεράντι του ξεπλήματος, γιατί αν δεν υπάρχει ξέπλυμα δεν υπάρχει Παναμά. Και από την άλλη στα πλαίσια της ανείχνευσης αυτών των δραστηριοτήτων μπορούμε να φέρουμε στην δημοσιότητα αυτούς οι οποίοι διαμεσολαβούν όπως σας είπα Ουάλα στα αραβικά. Ε, επειδή δεν υπάρχουν ανοιχτά σύνορα εκεί υπάρχει ένα σύστημα αντισταθμίσεων. Υπάρχουν επίσης οι ψευδείς τιμολογήσεις Και επίσης έχει σημασία στην ουσία είναι κάποιες ψευδεπίγραφες εμπορικές δραστηριότητες που επιτρέπουν όχι μόνο την αντιστάθμιση αλλά επιτρέπουν τη μεταφορά κερδών στο εξωτερικό. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν να έρθουν στην επιφάνεια αυτές οι παράνομες δραστηριότητες και να εντοπίσουμε και αυτούς οι οποίοι διαμεσολαβούν κάθε φορά. Ε, ψάξτε στο Google, πείτε ε, φορολογικός παράδεισος. Δεν θα σας μιλήσουν για τα Panama Papers. Έχετε 150 διαφημίσεις, ε, τραπέζες, ελβετικές και άλλες που θα σας επιτρέψουν να γλιτώσετε φόρους. Αυτή εξακολουθεί και τώρα να είναι η τάση. Πρέπει λοιπόν να εντοπίσουμε τα πρόσωπα αυτά. Πέμπτον, δέκα δευτερόλεπτα ακόμα. θα πρέπει με κριτήρια πιο διευρυμένα να ορίσουμε τι είναι φορολογικός παράδεισος και να φτιάξουμε νέους καταλόγους μη επαναλαμβάνοντας τα λάθη που είχαν κάνει οι προηγούμενες ομάδες έρευνας. Και στρέφουμε εδώ στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Οκτωβρίου του 2013 για τη διαφθορά. Είχατε κάνει μια εξαιρετική δουλειά, το οποίο πέταξαν στα σκουπίδια τα κράτη-μέλη. Εσείς είχατε προτείνει μέτρα τα οποία δεν ακολουθήθηκαν από τα κράτη-μέλη και θα έλεγα σε συνεννόηση με την Παγκόσμια Τράπεζα και το Δέλτα Νιτάφ είχατε προτείνει να γίνει κατανοητό ότι σε επίπεδο αριθματικό είναι βασικό σε παγκόσμιο επίπεδο να εννοήσουμε τις συνέπειες της καταστροφής της οικονομικής εγκληματικότητας έχουμε να κάνουμε με ε, μια θα έλεγα χωρίς προηγούμενη κατάσταση, με ένα συμβάν απερίγραπτο ε, και θα πρέπει να υπάρξει πολιτική ανταπόδοση εις βάρος των χωρών που θα εντοπιστούν στη διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστούμε Μίσελ Έχετε λοιπόν ε, μεγάλη εμπειρία και θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Νάουλη να πάρει το λόγο τελευταίος από το πάνελ μας από την Ειδική Υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος από τη Βορεια Ιρλανδία Βεσφαλία. Πείτε μας λοιπόν τη δική σας παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη συντομία τι κάνουμε ως ε, ερευνητέ στην υπηρεσία μας. Καταρχάς, ε, η ομάδα μας στην ε, Βορειοειρνανία Βεσφαλιά, της οποίας και ηγούμε, είναι καινούργια από τον Φεβρουάριο του 2015. Ομάδα ερεύνησης οικονομικού εγκλήματος και ο βασικός λόγος ύπαρξής της είναι η στενή σχέση της φορολογικής απάτης με άλλες απάτες γενικής εγκληματικότητας, είτε πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα ή άλλα οικονομικά εγκλήματα, διάφορα απάτη κτλ. Η φορολογική φοροαποφυγή επίσης συνδέεται σε πολλές περιπτώσεις, όπως έχουμε διαπιστώσει τελευταία, και με την τρομοκρατία. Για να βρούμε λοιπόν μια ευρεία προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις έρευνες και να έχουμε και δυνατότητε να εφαρμόσουμε τον νόμο με τους αστυνομικούς. Δημιουργήσαμε λοιπόν την ομάδα αυτή. Ε, μία έρευνα είναι η έρευνα Κανάλ, όπως το ονομάζουμε στα τέλη του 2013, η Βόρεια Ρενανία Βεσφαλία και οι οικονομικές υπηρεσίες μέσω των υπαλλήλων της από το Βούπερταλ έλαβαν πληροφορίες από έναν πληροφοριοδότη. Τις αγόρασαν τις πληροφορίες αυτές. Αυτές οι πληροφορίες φυσικά δεν ε, είναι αντίστοιχες των εγγράφων του Παναμά. Με τα έγγραφα του Παναμά εννοούμε τη δημοσίευση των δεδομένων εκείνων που έλαβε το ICIJ. Τα δικά μας τα δεδομένα, τι τα συνδέει με τα Panama Papers, το γεγονός ότι η δημιουργία τέτοιων εταιριών ε, offshore έγινε μέσα από την ε, εταιρεία Mossack Fonseca. Τα δεδομένα λοιπόν έχουν να κάνουν με την ίδρυση και την απόκτηση τέτοιων εταιριών offshore και σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με τις εταιρείε αυτές. Συγκεκριμένα τώρα. Βλέπουμε στα έγγραφα τα οποία έχουμε ότι το πιστοποιητικό ίδρυση των εταιριών, διάφορα πιστοποιητικά για αποφάσεις, τα πρακτικά των ε, συνεδριάσεων του Προεδρείου, εσωτερικά έγγραφα, πλήρη εξούσια. Εκεί αναφέρεται και ο δικαιούχος ε, και ο κάτοχος. Έχουμε το Μητρό των Μετόχων, τις ε, λογαριασμούς για την ίδρυση και τα τρέχοντα τέλη, ε, γιατί οι συντρέχονται αυτές οι εταιρείε. Έχουμε επίσης ε, πληροφορίες background για τις απομονωμένες εταιρείε και email επίσης μεταξύ των τραπεζών, των διαχειριστών των περιουσιών και της εταιρείας Mossack Fonseca δεν περιλαμβάνονται άλλοι τραπεζικοί λογαριασμοί και το υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασμών. Από τα στοιχεία λοιπόν αυτά προκύπτουν κάποια απορίσματα. Το όνομα του beneficial owner, του ιδιοκτήτη, το όνομα της ε, και η έδρα της εταιρείας offshore Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλες οι εταιρείε που έχουν ιδρυθεί μέσα τη Mossack Fonseca έχουν έδρα στον Παναμά. Όχι, και στι Αιχέλε και στα Κέιμαν κτλ. Η Mossack Fonseca είναι μια εταιρεία με 44, γραφεία που δραστηριοποιείται παγκοσμίω και έχει ιδρύσει εταιρείε σε όλε τι περιοχέ του κόσμου, όχι μόνο στον Παναμά. Και η έδρα δεν σημαίνει ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Φονσέκα ε, βρίσκονται στα νησιά Κέιμαν. Μπορεί να βρίσκονται και στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα ονόματα των τραπεζών, των διαχειριστών κτλ. και των υπαλλήλων. Εδώ έχουμε ένα σημαντικό στοιχείο ε, κρύβονται τα ονόματα των ατόμων αυτών. Και εδώ βλέπουμε ποιοι έχουν δραστηριοποιηθεί πραγματικά πως ε, Θα πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση την οποία να έχουμε παρατηρήσει όπου το beneficial owner, ο ιδιοκτήτης αυτός, είχε ίδιος επαφή με την εταιρεία. Αυτό πάντα συνέβαινε μέσω τραπεζών, υπαλλήλων, διάφορων χρηματοπιστωτικών πάροχων υπηρεσιών και το κόστος για την ίδρυση των εταιριών δεν τιμολογήθηκε κατευθείαν στην εταιρεία Φονσέκα. Πάντα μέσω τρίτων. Αν μία τράπεζα ζητούσε, για παράδειγμα, για τους, για τους πελάτες της ε, την ίδρυση μιας εταιρείας ε, offshore, ο πελάτης είχε επαφή μόνο με την τράπεζα αυτή. Αν ε, ο πελάτης άλλαζε τράπεζα, διαγραφόταν και η εταιρεία offshore. Η χρήση δηλαδή της ίδρυσης της εταιρείας συνδεόταν πάντα με ένα συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό σε μια συγκεκριμένη τράπεζα. Και όντως, αυτό το γνωρίζουμε, η δημοσιότητα και οι αρχές δεν μπορούσαν να διαπιστώσουν ποιος είναι πραγματικός ιδιοκτήτης. Και αυτό το πληρεξούσιο είναι ένα ιστορικό έγγραφο, το οποίο είναι γνωστό σε τρία μόνο άτομα. Ο ιδιοκτήτης, το γραφείο που δουλεύει στην Φοντσέκα και η τράπεζα ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Κανείς άλλος δεν είναι ενήμερος για το έγγραφο αυτό. Για μας λοιπόν, όταν ε, λάβαμε τα στοιχεία αυτά, ρωτηθήκαμε για ποιους σκοπούς μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς μια εταιρεία offshore, τι σκοπούς εξυπηρετεί και για... αυτό που είναι επίσης σαφές είναι το εξής ότι οι εταιρείε ε, offshore μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα βρωμικού χρήματος, ε, για την νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητε και για φορολογική φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή τώρα. Κατά 90% αποτέλεσε το ποινικό αδίκημα το οποίο κρυβόταν στις προκειμένες περιπτώσεις πίσω από τη δημιουργία τέτοιων offshore οι έρευνες, και ήταν εκτενέστατες οι έρευνες αυτές, τις ε, συνδέσαμε σε 524 ε, Γερμανούς πολίτες και με πάνω από 50 τράπεζες. Η υπόκτη ήταν η, η υπαλλήλη της Φονσέκα ε, για φορο διαφυγή. Και τα άτομα και οι υπάλληλοι οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην τράπεζα ή στο χρηματοπιστωτικό τρέμα. Και ο ιδιοκτήτης λόγω α, νομιμοποίησης παράνομων εισόδων από παράνομες ή για φοροδιαφυγή. Και έγιναν ε, έρευνες από το, την εισαγγελία της Κολονίας και από την εισαγγελία της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των ερευνών, ορίσαμε κάποιους στόχους σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των ερευνών. Ποινική καταδίκη, ε, επιβολή καταβολής των φόρων και κατάσχεση ενδεχομένω της διευθυνσίας και ενδεχομένως ε, ποινές ε, στις τράπεζες και στα χρηματοπιστωτικά εντρήματα. Γι' αυτό λοιπόν ε, αυτό πρέπει να γίνει μέσω διοικητικού δικαίου στη Γερμανία και φυσικά επιβολή κυρώσεων και στα φυσικά πρόσωπα. Στις έρευνες μας λοιπόν εστιαστήκαμε κυρίως στα άτομα εκείνα και τις υπηρεσίες εκείνες σε όλα τα επίπεδα που μπορούσαμε να βρούμε στο εσωτερικό, για παράδειγμα τις μητρικές εταιρείε γερμανικών τραπεζών με στο Λουξεμβούργο. Οι πάλι των τραπεζών, εφόσον είχαν τόπο κατοικίας ή τόπο άσκησης επαγγέλματος στη Γερμανία. Και όπως σας είπα, στο 90% των περιπτώσεων πρόκειται για φοροδιαφυγή και συνδρομή σε φοροδιαφυγή. Ένα βασικό κίνητρο σε πολλές περιπτώσεις για τις εταιρείε offshore ήταν η εταιρεία, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τα τελενιακά τέλη, εφόσον πρόκειται για Ευρωπαίο πολίτη και υποχρέωση καταβολής τέτοιων τελών. και έτσι μεταφέρα τον αναλογισμό σε εταιρεία offshore για μη καταβολή των τελών αυτών. Άρα, βασικό στόχος ήταν ε, να υποσκελιστεί αυτή η οδηγία. Και έτσι συνολικά πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η αρρωγή για τη φοροδιαφυγή, η οποία διαπιστώνεται και από άλλες τραπεζικές έρευνε, αποτελεί μια συστημική μορφή οικονομικού εγκλήματος. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να κλείσω την παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε μάθει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα από αυτά που είπατε, <clears throat> αλλά έχουμε και ένα πρόβλημα πίεσης χρόνου. Έχουμε χρόνο μονάχα μέχρι τις 6.30, ε, 45 λεπτά δεν κάνω λάθος. Έχουμε ένα μακρύ κατάλογο ομιλητών. Σας παρακαλώ να έχουμε χρονοθυρίδες τριών λεπτών. Ένα λεπτό ερώτηση, δύο λεπτά απάντηση, όταν αυτό είναι δυνατό. Ακόμα και ο κύριος ε, Μισελ ως ε, πρώην Υπουργός Εξωτερικών θα το αποδεχτεί πιστεύω. Ο κύριος Λούκε είναι ο πρώτος ομιλητής. Δεν συμφωνώ με αυτό κύριε Πρόεδρε, έχουμε συζητήσει ότι έχουμε το δικαίωμα να θέσουμε και συμπληρωματικά ερωτήματα σε αυτή την Επιτροπή. Εσείς μας περιορίσετε τώρα το χρόνο ομιλίας. δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί αλλιώ θα τελειώσει η συνεδρία και θα έχουν μιλήσει μονάχα οι συνάδελφοι. Έχουμε σαφείς ε, κανόνε, έχουμε και του διευνήσεις οι οποίοι πρέπει να σταματήσουν να δουλεύουν κάποια στιγμή. Εγώ κάνω μια πρόταση να περιστείλετε το χρόνο και ίσω κάποιοι μπορούν να θέσουν σύντομα ερωτήματα για να μην καθυστερήσουμε. Κύριο Σκόφον, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Για τον Φιλίπ Ντεκοστέρ σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Μία από τις προτάσεις σας είναι ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή υπηρεσία καταστολής των ευρωπαϊκών παραβάσεων για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Έχετε κάποια πρόταση. Αν είχαμε μια τέτοια ευρωπαϊκή υπηρεσία συλλογής πληροφοριών για τη φυρολογία θα λειτουργούσε καλύτερα. Είπατε ότι υπάρχουν ε, αρκετές περιπτώσεις Βέλγων στα Panama Papers. Ζητήσατε πληροφορίες από τον Παναμά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Και τέλος, για τον κύριο Ναουλίνα, η μέθοδος την οποία χρησιμοποιήσατε, αγορά πληροφοριών από πληροφοριοδότες, το κάνουν και οι Δανείοι αυτό. Σας βοήθησε αυτό, το συστήνετε και σε άλλες χώρες. Αγορά δηλαδή στοιχείων. Σας ευχαριστώ για το σύντομο των ερωτήσεων. Ο πρόεδρος Κώστερ έχει το λόγο. E Απαντήσω λίγο σύντομα, λέει ο κύριος Δεκώστερ είναι κάτι το οποίο έχει τεθεί επιτάπητος εδώ και πολύ καιρό. Δεν χρειαζόμαστε πολλά λεφτά, δεν χρειαζόμαστε νέα κτίρια και νέες υπηρεσίες. Θέλουμε απλώς το θάρρος να κάτσουμε και να συζητήσουμε και να αναλύσουμε αυτό που βρίσκεται μπροστά από τη μύτη μας εδώ και πολύ καιρό. Και αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα που μπορούμε να αντλήσουμε σε σχέση με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. <clears throat> Πρέπει να έχουμε μια κοινή ομάδα έρευνας από, τους, ε, από τις μονάδες ε, συλλογής πληροφοριών για τα χρηματοπιστωτικά. Και εδώ υπάρχει συνεργασία ήδη με άλλες ε, υπηρεσίες, <clears throat> αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όχι μόνο τι είναι χρήσιμο για μα και να περιμένουμε, αλλά και τι είναι χρήσιμο για του συναδέλφου μα και όχι να περιμένουμε να μα ζητήσουν κάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτέ τι 97 περιπτώσει, τίποτα απολύτω. Εξαρτάται από τον εισαγγελέα του Παναμά. Θα απαντήσει στο ερώτημά μου. Θα απαντήσει η μονάδα χρηματοπιστωτικών πληροφοριών αυτό το ερώτημα. Τι θα κάνετε αλλιώ, τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε. Είναι κάτι το οποίο δεν μα ικανοποιεί. Κύριο Νάουλιν, λέει ο πρόεδρο. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι <clears throat> σε παγκόσμιο επίπεδο τα ποινικά συστήματα ε, μάλλον μπορεί μέσα σε αυτά τα συστήματα που έχουν να κάνουν με το έγκλημα, ε, με το έγκλημα ότι μπορεί να ξέρει κανείς να καταλάβει κανείς κάτι όταν έχει πληροφορίες εκ των έσω. Δεν υπάρχει αλτρουιστική αντιμετώπιση μεταξύ των αρχών υπάρχει πάντα ένα βασικό ερώτημα. Το θέμα των χρημάτων και το θέμα επίσης της, πληρο... της προστασίας των πληροφοριοδοτών. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα σύστημα προστασίας των καταγγελόντων, των whistleblower, που θα πρέπει να σκεφτούμε μέχρι πού πρέπει να φτάνει αυτό, αλλά αυτό πρέπει να γίνει σε νομοθετικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μισελ ο οποίος ε, αντικαθιστά τον κύριο Γιατσέκ. Ναι κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντεκοστέρ, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πριν από τις αποκαλύψεις των Panama Papers, είχατε στο παρελθόν γνώσεις ή υποψίες ότι μπορούσε να συμβαίνει κάτι. Είχατε στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να σας οδηγήσουν στο να προβλέψετε το θέμα του Παναμά. Εάν ναι, γιατί δεν κρούσατε το κόδωνο του κινδύνου προηγουμένως. Και γιατί δεν έγιναν έρευνε πριν από την αποκάλυψη των Panama Papers. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Τι περιμένετε από την Europol, γιατί είχα την εντύπωση από την ε, απάντησή σας στην γραπτή, στις γραπτές ερωτήσεις, ότι θεωρήσατε ότι δεν είσαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένο από τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόντουσαν οι, οι μονάδες χρηματοπιστωτικών πληροφοριών με την Europol. Επίσης, εγώ κατανοώ την αγανάκτησή σας, αλλά δεν ε, συμμερίζομαι την πικρία σας. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι. Υπάρχει ένα στοιχείο για το οποίο θα ήθελα να έχω την άποψή σας. Εγώ είχα την ευκαιρία να αναφέρω αυτό. Πιστεύω αυτό, αυτοί που ονομάζετε εσείς διευκολυντές δεν είναι ακριβώς το στόχαστρο ακόμα. Έχω την εντύπωση ότι αυτοί ξεφεύγουν από την αγανάκτησή σας, ξεφεύγουν από τις έρευνές σας και αυτό με σοκάρει. Γι' αυτό θέλω να έχω την άποψή σας για το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των διευκολυντών, γιατί χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν δυνατό. Δεν θέλω λοιπόν να ξεφύγουν από την ε, ε, δίωξη και από την κρίση σας. Ευχαριστώ κύριε Μισελ. Δύο λεπτά μιλήσατε. Μέχρι στιγμής κανείς δεν κράτησε απόλυτα το χρόνο αυτό και σε άλλες ακρόασεις. Δίνω το λόγο στον κύριο Κώστερ. Κύριε θα σας απαντήσω με αριθμούς. Τον Ιανουάριο του 2014 έκθεση του Δέλτα Νιτάφη για τον Παναμά για την καταπολέμηση του ξεπλήματος, την χρηματοδότηση της δημοκρατίας ε, και την υπηρεσία συλλογής οικονομικών πληροφοριών. Λέει το Δελτανιτάφ ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, έχει περιορισμένους πόρους η υπηρεσία, καθυστερεί, δεν κάνει δουλειά. Τον Οκτώβριο το 2014 το Βέλγιο στην ομάδα ΕΓΜΟ ε, λέει ότι με τον Παναμά έχουμε πρόβλημα, μπορούμε να βοηθήσουμε, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει συνεργασία. Τον Ιανουάριο του 2016 το καφί πηγαίνει επί τόπου, τα λύνουν όλα, πηγαίνουν επί τόπου, τα βρίσκουν όλα καλά. Το Φεβρουάριο του 2016 ο Παναμά συνεργάζεται και τον Μάρτιο τον Απρίλιο μάλλον του 16 οι δημοσιογράφοι τα βγάζουν όλα στην επιφάνεια. Συνεπώς λοιπόν γι' αυτό πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στην υπηρεσία συλλογής στοιχείων, πληροφοριών και τη Europol. Η δική μου υπηρεσία είναι μια διοικητική υπηρεσία. Στο ΣΕΡΕΦ στο Λουξεμβούργο είναι δικαστική. Η Europol είναι αστυνομική. Αν τώρα αρχίζουμε να φέρνουμε σε αντίθεση τα μοντέλα μας, γιατί οι μένοι είναι αστυνομικοί, οι άλλοι είναι δικαστές κτλ, αυτό είναι γελίο. Εμείς ξεπεράσαμε τις διαφορές και θα πρέπει να κάνουν το ίδιο και οι άλλοι. Μοντανιέ και μεταμπλάζ. Ο κύριος Κλάις, απαντώντας τον κύριο Μισελ σχετικά με τους διαμεσολαβητές. Νομίζω ότι αν μπορέσουμε να παρέμβουμε εκεί θα στερήσουμε τη μαφία από τους ανθρώπους που τους προστατεύουν και θυμηθείτε και το έργο με τον Τόμ Κρούζ όπου λέει ότι για να χτυπήσεις τη μάφια χτυπάς τους δικηγόρους της. Λοιπόν, ξέρετε, πηγαίνετε σε μια έκθεση στο Χάιζελ και για επιχειρηματίες και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σας προτείνουν τέτοιου είδους φορολογικές διευκολύνσεις. Υπάρχει σαλόνι πρέτα πόρτε της φορολογικής απάτης από τη Γενέβη μέχρι τη Μόσχα. Εταιρείε offshore, Panama Papers και η πρώτη συνάντηση είχε γίνει στο Grand Palais στο Παρίσι το 2000 και ε, χρηματοδοτήθηκε από την Ένωση, από τον UBS, από τη Mercedes και από την Price and Waterhouse. Συνεπώς λοιπόν, αυτοί οι οποίοι μπορούν δωρεάν να καταγγέλουν και να δίνουν τέτοια στοιχεία, ε, ήδη στη Γερμανία αγόρασαν στοιχεία από το Liechtenstein, από συγκεκριμένους ε, ε υπαλλήλους τραπεζών. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα βέβαια, γιατί σε επίπεδο ποινικού αυτό θεωρείται προϊόν διαφθοράς. Θα σας ευχαριστώ επόμενος για το ΕΛΚΑ, ο κύριος Νίτερ Μάια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα αυτά που μάθαμε για τα έγγραφα του Παναμά, φαντάζομαι ότι συνδέονται σε κάποιο βαθμό και με το παρελθόν και μεταξύ έχει αλλάξει μεγάλο τμήματα της νομοθεσίας. Άρα ερωτώ, Αυτές οι αλλαγές σε τι βαθμό έχουν βελτιώσει την κατάσταση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος και άλλες τέτοιες νομοθετικές προσπάθειες. Και με ένα βλέμμα προς το μέλλον ρωτήσω το εξής. Ε, προβλέπετε νέα αναθεώρηση της νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος και τα πρότυπα του ΆΣΑ και θα ξεκινήσουν όλα αυτά από το χρόνο. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν όλα αυτά. Θα μειώσουν ε, απλά το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Πριν δώσουμε το λόγο για να απαντήσουν οι πανελίστες, να δώσω το λόγο στον κύριο Μοντουαγέ. Μοντανιέ. Κοιτάξτε, για, τις, για τους επόπτες ε, και τους ελεγκτές, τους προληπτικούς ελεγκτές, των πιστοτικών ε, ε, συναλλαγών, των τραπεζικών συναλλαγών. Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε αν ε, πράγματι μπορούν να ελέγξουν την προέλευση των κονδυλίων, των ποσών. Και αν υπάρχουν αμφιβολίες τότε θα πρέπει να καταθέτουν την αναφορά υποψίας στις υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών. Κάθε φορά που υπάρχουν βελτιώσεις και ήδη η τέταρτη οδηγία ενισχύει θα έλεγα τις προσδοκίες που έχουν οι διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες. Αυτό επιτρέπει τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος. Από την άλλη κάθε φορά που υπάρχει μια άλλη χώρα όπου οι νομοθετικές ρυθμίσεις επιτρέπουν να αποκριβούν κάποια στοιχεία, τότε είναι προφανές ότι το σύστημα δεν θα λειτουργήσει σωστά νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια να συλλέγουμε στοιχεία για τις πρακτικές που ακολουθούν οι διάφορες ελεγκτικές υπηρεσίες. Δεν υπάρχει αν θέλετε η ενιαία συνταγή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Μπορούμε ίσως να καταστήλουμε κάπως το φαινόμενο αλλά όχι να το εξαφανίσουμε. Ευχαριστώ. Θέλει να πάρει το λόγο για να συμπληρώσει κάτι, ο κύριος Κλάης. Κοιτάξτε, τα νομοθετικά, νομοθετικά όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, λαμβάνονται και χρησιμοποιούνται αναχώρα. χώρα. Εμείς ε, επιβάλαμε στους επαγγελματίες, αν θέλετε, ε, του χώρου να δηλώνουν τα στοιχεία σχετικά με τους πελάτες τους αλλά πολύ συχνά γίνονται έλεγχοι και στις υπηρεσίες ορκωτών λογιστών, αλλά όχι σε επίπεδο δικηγόρων. Εγώ όταν ψάχνω ως δικηγόρου σαν παράδειγμα να βρω στοιχεία και καταλόγους πελατών κτλ δεν βρίσκω τίποτα. Το πραγματικό πρόβλημα λοιπόν είναι η έλλειψη μέσων που χαρακτηρίζει τα δικαστικά συστήματα. Έχουμε μέσα, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα και σε επίπεδο αστυνομικό και σε επίπεδο δικαστικό. Και αυτό είναι καταστροφικό σαν φαινόμενο. Έχετε το λόγο. Σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές τροποποίησεις, πιστεύω ότι προς τη σωστή κατεύθυνση πηγαίνουν. Αλλά εγώ ως ερευνητής μόνο στο παρόν μπορώ να αναφερθώ, δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει στο μέλλον και ποιες θα είναι οι συνέπειες. ό,τι αφορά όμως τα νομοθετικά, πιστεύω ότι υπάρχουν ε, κάποια πράγματα που με απασχολούν ιδιαίτερα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό λοιπόν το, ε, περιλαμβάνει το εξή. Θεωρώ ότι χρειάζεται μία ένα σαφή ορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το τι αποτελεί ε, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και μια εναρμόνιση σε ό,τι αφορά το ποινικό μήτρο στην Ευρώπη. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ τη νομική συνεργασία σε διμερέ επίπεδο, που σε πολλέ περιπτώσει δεν είναι αρκετά απλή σε διμερέ επίπεδο και πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι και να προβλέπεται σε όλες τις ε, χώρες ότι η φόρο διαφυγή αποτελεί ξεπλήρωμα μαύρων χρήματος. Αυτό δεν είναι εγγυάται σε όλες τις χώρες. Ότι αποτελεί αδίκημα. Δεν είναι πάντα αδίκημα. Και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και καλύτερη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ενδεχομένω χρηματοδοτούνται με παράνομο τρόπο. Αυτό θα μπορούσε να ρυθμιστεί πραγματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Σημειώνουμε τι προτάσει σα. Ο κύριο Ουκ Μπαγιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όπως είπατε και εσείς κύριε Ντεκοστέρ, οι διευκολυντές είναι πάντα πάρα πολύ ενεργοί και είναι αυτοί που παίζουν τον ε, απαραίτητο ρόλο. Έχετε την εντύπωση ότι υπάρχει και διαφορά αντιμετώπισης διαφορετικών ε, επαγγελμάτων και πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε την ε, νομοθεσία. Χαίρομαι λοιπόν <clears throat> ότι θα ακούσουμε και αυτούς τους διευκολυντές οι οποίοι λένε ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα, εμείς εφαρμόσουμε την νομοθεσία μονάχα θα ήθελα να έχω και τη δική σας άποψη ως εργασόμενου επί των θεμάτων αυτών, πώς πάντα πάμε τα μεταξύ κρατών μελών και των ευρωπαϊκών οργάνων. Ακούσαμε την άποψη των θεσμών, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη για το θέμα αυτό και το τελευταίο μου ερώτημα, το οποίο είναι ίσως ευρύτερο. Αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ξέπλυμα χρημάτων, ότι πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Είδαμε τις τελευταίες αλλά τι μέτρα ακόμα μπορούμε να πάρουμε για να σα βοηθήσουμε περισσότερο στο έργο σα. Ευχαριστώ. Merci, Ποιος θα ήθελε να απαντήσει, ο πρόεδρος Δεκοστέρ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Με λίγου αριθμού εδώ μιλήσαμε για φορολογικέ απάτε και αναφερθήκατε στην συνεργασία με τις υπόλοιπες χώρες. Το 2015 ασχοληθήκαμε και μεταφέραμε στις δικαστικές αρχές οκτώ φακέλους φορολογικής σοβαρής οργανωμένης απάτης που δεν ήταν σχετική με το Βέλγιο. Η απάτη αυτή αφορούσε το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης είχαμε και για την Πολωνία, τη Σιγκαπούρη και τη Μαδαγασκάρη. Τώρα, για... έχουμε ένα φάκελο για Βέλγους στο εξωτερικό και το στοιχείο μας το έδωσε στο Λουξεμβούργο. Και έχουμε και άλλο ένα που μας έδωσε στοιχείο το Χονγκ Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι δεν έχουμε περιθώρια. Σε επίπεδο φορολογικής απάτης πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Δεν είναι θέμα συνεργασίας. Εγώ μπορώ να συνεργάζομαι με τους συναδέλφους του Κρεφά όταν αναφέρομαι ε, σε φορολογικές απάτες εις βάρος του γαλλικού κράτους. Όταν όμως τους ζητάω τα στοιχεία ε, των απαταιώνων των Βέλγων που από τη Γαλλία κοροϊδεύουν το Βέλγιο δεν μου λένε τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ορίσουμε με διαφορετικό τρόπο τις απάτες. Ένα άλλο παράδειγμα τώρα ε, σε συνεργασία με το Κέντρο Συλλογής Οικονομικών Πληροφοριών του Λουξεμβούργου. Ε, ψευ, ψευδής φορολογική απάτη, δηλαδή ε, γύρω στα 100 εκατομμύρια πηγαίνουν στο Λουξεμβούργο, προέρχονται από μια πτωχευμένη εταιρεία εδώ και 10 χρόνια, με πολλούς που έμειναν στο δρόμο γιατί έκλεισε η εταιρεία και μιας και το εγκλη... η ομολογημένη αμαρτία είναι μισή αμαρτία, λένε ότι τώρα μια και κάναμε μια απάτη θέλουμε να την επανορθώσουμε με μικρό κόστος βέβαια. Στην ουσία έχουμε να κάνουμε με ένα διπλό μηχανισμό. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι για να τα δούμε τα πράγματα πιο θετικά. Έχουμε ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας στην Eurojust μαζί με την Europol Έχουμε αυτές τις κοινέ ομάδες έρευνας μετά από τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Αυτή είναι, μας δίνει τη δυνατότητα με μια συμφωνία των δικαστικών αρχών να μην περάσουμε με το πολύ βαρύ σύστημα των διεθνών επιτροπών ε, έρευνας και να έχουμε αμέσως συνεργασία. Κάποια στιγμή είχα ζητήσει μια ε, έρευνα κατοίκων στην Βασοβία η οποία εφαρμόστηκε αμέσως. Η Eurojust μας δίνει και πολύ καλό υλικό μαζί με μεταφραστές για τις διεθνείς ε, συμφωνίες, καλύπτει τις, ε, το κόστος των ερευνών για άλλες χώρες όπως είναι το Μαρόκο. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τις χώρες ΜΕΡ. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς επιτροπές έρευνας υπάρχει αυτό το σύστημα <clears throat> το οποίο λειτουργεί. Υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη η οποία δεν απαντάει καθόλου. Ε, έχουμε καταφέρει σε διεθνές επίπεδο να έχουμε συνεργασία με θαυμάσια με χώρες ε, όπως και το Πακιστάν, η Ρωσία και άλλες περιπτώσεις που δεν είχαμε καμία απάντηση. Ευχαριστώ, Διαπρόεδρος, ο Μπέντ Λούκε για το, για, ε, το ECR. Μία ερώτηση προς τον κύριο Μιλήσατε για τη σημασία των ε, συμβούλων στις τράπεζες, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ό,τι αφορά τη σύνδεση και με τη Μονσέκ Φονσέκα και σε ό,τι αφορά ε, την παροχή συμβουλών προς τους ε, ιδιοκτήτες των εταιριών. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως για να μην διώκουμε ποινικά τα μικρά ψάρια, αλλά τους μεγάλους υπέτειους, μεγάλες εταιρείε στις γραπτές απαντήσεις αναφέρατε ότι 95% των περιπτώσεων που ερευνείται είναι στο Λουξεμβούργο και είναι θηγατρικές γερμανικών τραπεζών. Άρα οι αποφάσεις λαμβάνονται σε υψηλό επίπεδο στις τράπεζες για να εγκαταστήσουν τις θηγατρικές στο Λουξεμβούργο. Και άρα ερωτώ, η ποινική δίωξη στρέφεται και κατά ατόμων που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και φέρνουν ευθύνη ε, στις ε, γερμανικές τράπεζες για τις δομές αυτές. Και ρωτώ λοιπόν, τι χρονική πίεση αντιμετωπίζεται λόγω του κινδύνου ε, χρονικών περιορισμών παραγραφής σε ό,τι αφορά δηλαδή τη δυνατότητα επιβολής κυριώσεων λόγω του κινδύνου παραγραφής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε και για απάντηση τώρα. Φυσικά, καταρχάς, ε, εντοπίζουμε τους συμβούλους της τράπεζας και κοιτάμε ποιος είναι σε άμεση επαφή με τον ε, πελάτη και είναι γνωστό ότι ένας ε, υπάλληλο ο οποίος δραστηριοποιείται ως σύμβουλος δεν είναι τυχαίο σε μια τράπεζα και φυσικά προσπαθούμε να δούμε και τις ευθύνες ανά επίπεδο και ανάλογα με την ιεραρχία. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να βρούμε και κάποιο συγκεκριμένη ενδείξη για κάθε κατηγορία. Και εδώ δυσκολεύουν τα πράγματα κάπω. Το θέμα είναι το εξή. Οι γερμανικέ τράπεζε δεν έχουν μόνο θηγατρικέ στο Λουξεμβούργο, αλλά αυτέ που είναι στο Λουξεμβούργο ουσιαστικά είναι κανονικέ θηγατρικέ ε, εταιρείε. Και έχουν και κανονικέ δραστηριότητε, όπω οι κανονικέ τράπεζε. Και σε ό,τι αφορά τα στοιχεία μας, εστιαζόμαστε μεν στο Λουξεμβούργο, αλλά δεν είναι ότι οι τράπεζες, οι θεατρικές αυτές, ε, ιδρύονται προς, προς την κατεύθυνση αυτή και για τον σκοπό αυτό. Πάντα ε, ανέκαθεν υπήρχαν αυτές οι τράπεζες και δραστηριοποιούνταν σε κανονικές δραστηριότητες. Και φυσικά εξυπηρετούν όχι μόνο αυτούς που είναι στο Λουξεμβούργο, αλλά και οι Γερμανούς. Και κοιτώντα τα φυσικά πρόσωπα, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα φυσικά πρόσωπα, επειδή δεν υπάρχει συγκεκριμένο δίκαιο που να μπορούμε να εφαρμόσουμε κατά φυσικών προσώπων, ουσιαστικά τιμωρούμε το νομικό πρόσωπο. Τέτοια τα θέματα ε, παραγραφής δεν έχουμε. Και έχουμε μία δεκαετή τέτοια περίοδο παραγραφής σε μία περίπτωση που είχαμε κάποια τέτοια ζητήματα, ε, έχουμε κάνει κάποια βήματα για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο τη παραγραφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαγατσούντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για σε όλου σα. Λαμβάνουμε υπόψη τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μα δώσατε. Εγώ ε, πρόκειται να έρθει ε, ένας... Υπήρξαν και πολλοί φόροι άλλοι οι οποίοι έλαβαν το λόγο ενώπιον μας. Εν πάση περιπτώσει ο κατάλογος των φορολογικών παραδείσων είναι κάτι που είναι δύσκολο να έχουμε χωρίς να έχουμε σαφή κριτήρια. Δεν θα είναι εύκολο η κατά... κατάλογη αυτή λοιπόν να είναι αποτελεσματική. Μιλήσατε για τους διευκολυντές και τέθηκε αυτό το ερώτημα του πώς θα μπορέσουμε να παρεύουμε με πιο στεναρό τρόπο εναντίον αυτών που διευκολύνουν την ε, διαδικασία αυτή. Αυτό το οποίο έχουμε μάθει από τις διαρροές στα Panama Papers, θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο θεωρείτε ότι η οδηγία για τη λεύκανση χρημάτων είναι <clears throat> κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει πιο <clears throat> συστηματικά για να βρούμε του ενδιάμεσου, δηλαδή όπω κάνουμε και στην περίπτωση των, του ελέγχου τη τρομοκρατίας σε αεροπορικέ γραμμές, πώ μπορούμε να κάνουμε κάποιο screening για να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, εφόσον φυσικά υπάρχει πολιτική θέληση για κάτι τέτοιο. Θα ήθελα επίση να, να γνωρίσω την άποψή σα για την φορολογική αμνηστία, για τι φορολογικέ αμνηστίε που γίνονται. Στη δική μου χώρα αυτό έχει οδηγήσει σε μια κάποια ατιμορρησία και θέλουμε επίσης να αποφύγουμε κάθε είδους σφάλματα. Λέτε ότι τα πρότυπα είναι σωστά, αλλά δεν έχουμε υλικά και ανθρώπινα μέσα. Πέστε μας τι χρειάζεστε για να μπορέσετε να λύσετε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα ήθελε να απαντήσει από εσά πρώτος. Φορολογικές αμνηστίες και πού βρίσκεται αυτό, κύριος ε, ε, Μοντανιέ. Α, πρώτα, ας ξεκινήσουμε με το Βέλγιο. για το θέμα των ρυθμίσεων των φορολογικών. Ε, το γνωρίζουμε στο Βέλγιο, εμείς βρισκόμαστε στην τέταρτη τέτοια αντίστοιχη διαδικασία. Η πρώτη ήταν διαδικαστική, η δεύτερη και η τέταρτη ε, σημειώνονται από ένα σημαντικό ρόλο της υπηρεσίας μας, περίπλοκο όμως, που αντίθετα από ό,τι πιστεύει κανείς δεν μας εμποδίζει να δράσουμε. Εγώ εξέθεσα κάποιους φακέλους για το ξέπλυμα και για παράνομες ε, ε, πτωχεύσεις. Νομίζω ότι το σύστημα με δυσκολίες μπορεί να δουλέψει. Το να υπάρχουν ρυθμίσεις φορολογικές, αυτό είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει η κυβέρνηση. Αλλά να μην ρυθμίζονται αυτές οι διευθετήσεις υποφορολογικές για να ξεπλένεται χρήμα προϊόν εγκλήματος. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι ακόμα. Κύριος Νόιλιν. Νάουλιν. να σταθώ τώρα στο θέμα των συμβούλων. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είναι δύσκολο να αποδείξει κανείς τι ακριβώς κάνει ένας σύμβουλος αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι ε, υπάρχει μια υποχρέωση να δηλώνονται οι δραστηριότητε των ε, συμβούλων και επομένως να έχουμε την δυνατότητα τουλάχιστον από τις μεγάλες επιχειρήσεις να έχουμε γνώση για το ποιοι τους, ποιους συμβουλεύουν. Αυτό θα ήταν μια χρήσιμη λοιπόν πιστεύω ε, διάταξη. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάτι που είπαν και οι συνάδελφοι, ότι υπάρχουν κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να μπορούν να αρθούν, να εφαρμοστούν, συγγνώμη, και η εφαρμογή χρειάζεται πολλά χρήματα και πολύ χρόνο και προσπάθεια. Υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο, κυρίως ε, ο Φάμπιο Δημάση για την ΚΟΥΕΧ. Ναι, ναι, παρακαλώ. Είσαστε έτοιμος να απαντήσετε. Εγώ έλεγα ότι δεν είμαι σε θέση να μιλήσω για τις διαφετήσεις αυτές τις φορολογικές. Δεν είναι κάτι το οποίο εντάσσεται στις δικές μου αρμοδιότητες. Αυτό το οποίο όμως παρατηρούμε για μια ακόμη φορά είναι ότι η δικαιοσύνη μπορεί να καταδικάσει και άλλους ενδιαμέσους, όχι μόνο τράπεζες, συμβούλους, δικηγόρους, αλλά εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η τράπεζα να έχει κάνει τη δουλειά της και να έχει καταθέσει την λεγόμενη δήλωση υποψίας αν θέλετε. Εμείς πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο έλεγχος μιας ομάδας, ενός ομίλου, να γίνεται όχι μόνο στο εσωτερικό των εθνικών συνόρων. Και εδώ έρχεται και η αναθεώρηση της τέταρτης οδηγίας που θα μπορούσε να βελτιώσει τη συνεργασία καθιστώντας την πιο συστηματική και υποχρεωτική έτσι ώστε οι ελεγκτές μιας ομάδας ενός ομίλου επιχειρηματικού να συναντάτε και να συνομιλεί με τους επόπτες και τους ελεγκτές των υπολείπων εταιριών του ιδίου ομίλου. Γιατί από τη φύση τους πάρα πολλές από τις επιχειρήσεις που μας ενδιαφέρουν είναι πολυεθνικές, ντεμάζει. Ένα ερώτημα προς τον κύριο Νάουλιν. Ε, είναι πολύ θετικό το ότι, ότι έχετε αναφερθεί στην νομοθεσία. Έχουμε την οδηγία κατά της λεύκανσης χρημάτων, η οποία κατά την άποψή μου εξακολουθεί να έχει πάρα πολλά παραθυράκια, τα οποία θα πρέπει να κλείσουν αν θέλουμε να υπάρξει πραγματική ρύθμιση των θεμάτων αυτών. Εσείς μπορείτε να μου πείτε από τη δική σας εμπειρία γιατί δεν μπορεί μια εταιρεία να έχει ε, πληροφορίες για τους... Ε, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η έρευνα για τους τελικούς, για τους ε, τελικούς δικαιούχους. Υπάρχουν ε, όλες αυτές οι εταιρείες γραμματοκιβωτίου, οι οποίες υπάρχουν και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς βλέπετε όλη αυτή η προβληματική. Παρακαλώ. φοβάμαι ότι η φαντασία και η δημιουργικότητα αυτών οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα παραθυράκια είναι ανεξάντλητη. και όλες οι ευκαιρίες οι οποίες είναι δυνατόν να τύχουν εκμετάλλευση θα γίνουν. Δεν μπορεί κανείς να κάνει τον κόσμο καλύτερα, μπορεί να κάνει πιο στενό το πλαίσιο για παραβίαση. Βέβαια είναι όπως το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί κανείς να αποτρέψει όλες τις, όλα τα κόλπα τα οποία γίνονται. Είναι απαραίτητο όμως να θέσουμε τις επιχειρήσεις και τους παρόχους ε, υπηρεσιών ώστε στο βαθμό του δυνατού να έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους, ε, δι, για τους ε, δικαιούχους κτλ. Η Εύα Ζολή από τους πράσινους έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεκινώντας θα έλεγα ότι τα Panama Papers και τα τεράστια ποσά που γίνονται αντικείμενο διαχείρισης από τους φορολογικούς παραδείσους και που γνωρίζουμε από την Τράπεζα Διεθνών Ρυθμίσεων euh, για κανονισμών ε, είναι ανησυχητικά τα ύψη των ποσών αυτών. Να μας πει ο κύριος Μοντανιέ ε, σε ποιο βαθμό είναι πλεονέκτημα να μπορεί κανείς να ελέγξει προληπτικά τις τράπεζες της ασφάλειας και για τους τραπεζικούς κινδύνους και για τους κινδύνους από το ξέπλυμα χρήματος. Είναι δυνατό να καλύψετε όλους αυτούς τους τομείς ε, και τι κυρώσεις προβλέπετε για την Societe Generale και την BNP για τον αριθμό των επιχειρήσεων offshore που έχουν δημιουργηθεί και καταχωρηθεί από την Mossack Φονσέκα γιατί οι επιχειρήσεις αυτές κατά το 90% δυστυχώς η εμπειρία μας από τις αμερικανικές μελέτες δείχνει ότι έχουν εγκληματικούς στόχους. Ο κύριος Μοντανιέ. το πλεονέκτημα αν θέλετε του να έχει κανείς κάτω από το ίδιο καπέλο και την χρηματοπιστωτική ασφάλεια ενός κράτους και το θέμα του σεβασμού των γαλλικών και διεθνών κανόνων για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μας επιτρέπει να κρίνουμε για το εάν ή όχι έχουμε την δυνατότητα να κατανοήσουμε τη διάθεση ε, ε, ενός οργάνου όταν οργανώνει τις ελεγκτικές του δραστηριότητες. Το πεδίο είναι τεράστιο και στον τομέα των προληπτικό και στον τομέα του ξεπλήματος. Οι έρευνες που κάνουμε είναι πολύ μεγάλες, αλλά δεν μπορούμε να ελέγχουμε όλα τα, όλες τις, τα πιστοτικά ιδρύματα φυσικά συνεχώς και σε αιτήσια βάση. Σχετικά τώρα με τις ε, μεγάλες εταιρείες και τα μέσα offshore στο εξωτερικό. Δεν είναι από τη φύση τους παράνομα. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να επιβάλλουμε κυρώσεις στις τράπεζες είναι αν έχουν βγάλει χρήματα από τη Γαλλία με ασύμβατο προς τον γαλλικό νόμο τρόπο ή αν έχουν επίσης οργανώσει κάποιες δραστηριότητες στις θηγατρικές τους επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ασύμβατες είτε με το διεθνές δίκαιο είτε με την εθνική νομοθετική ρύθμιση. Είναι δύσκολο να το ελέγξουμε αυτό. Εμείς δεν είμαστε δικαστική αρχή και για κάποιες χώρες του εξωτερικού δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πράγματα επιτόπου γιατί δεν έχουμε ε, την δυνατότητα δυστυχώς να δούμε τι κάνουν εκεί οι γαλλικές τράπεζες, για αυτές μιλάω τώρα. Ε, πολλές αρχές από διάφορες χώρες ε, είπε ότι μπορείτε να δείτε τις επιχειρήσεις αυτές αλλά δεν έχει νόημα γιατί δεν θα σας δώσουμε τους, αρχι... τους υπευθύνους των λογαριασμών, τα ποσά που περνούν και τα κέρδη τους. Λοιπόν, εμείς ελέγχουμε την παραβίαση του γαλλικού δικαίου ή των τραπεζικών κανόνων που μπορεί να είναι κάτι το ανιχνεύσιμο. Δυστυχώς όμως, επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να πάμε στις συγκεκριμένες χώρες φορολογικούς παραδείσους. Σας ευχαριστώ και έχουμε άλλους δύο μιλητές στον κατάλογο των ομιλητών. Η ε, κυρία συγκεκριμενες χωρες φορολογικους παραδεισους σας ευχαριστω και εχουμε αλλους δυο μιλητες στον καταλογο των μιλητών. η κυρια ραμονοτο και η κυρία Αναλίζα και 20 δεύτερα ε, για όλες τις ερωτήσεις ε, την κυρία Γόμες. Ραμόνα. Ρωμάνα Βέρνερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. συντομία και μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση και για τους τρει ομιλητέ, αλλά ίσως πιο πολύ για τους πιο σχετικούς. Ε, τι πιστεύετε για τον τρέχοντα ορισμό των πολιτικώ εκτεθειμένων ατόμων, όπως περιγράφεται στην οδηγία για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματο. Είναι πολύ ευρύ, ο ορισμός, πολύ στενό ή σωστό Πολύ καλή ερώτηση. ποιο να ξεκινήσει, ο κύριο Προεδρο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσταθεί τίποτε στον ορισμό, αλλά αυτό που λείπει στην παρούσα είναι μια τεράστια βάση δεδομένων με όλα τα ονόματα όλων των ε, ε, υπετίων ε, μάλλον όλων των πολιτικών εκτεθειμένων ατόμων σε όλο τον κόσμο. Στη χώρα μου είναι εύκολο να ξέρουμε ποιο είναι ποιο. Αλλά όταν περνάμε τα σύνορα, τα πράγματα δυσκολεύουν κυρίω για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και νομίζω ότι εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει μια πρωτοβουλία για να δώσει μέσα και εργαλεία στους εμπλεκόμενους φορείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριο Κλέης, όχι. Ο κύριος Ναουλίν, όχι, ούτε αυτός επιθυμείται λόγο. Έχετε κάποια παρατηρήση να κάνετε. Είναι πολύ ευρύ ορισμό για μα. και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ελέγξουμε και να το πιστοποιήσουμε γιατί όντω δεν έχουμε κάποια βάση αναφοράς. Θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν βάσει των κριτηρίων να κάνουμε την σχετική έρευνα για το κατά πόσον τα χρηματοπιστικά ιδρύματα, τα ασφαλιστικά ιδρύματα όντω ε, καλύπτουν όλα τα άτομα τα εμπλεκόμενα. Και αυτό είναι πάντα προβληματικό για τον νομοθέτη για να υπάρχει σωστή αποδοτικότητα και να υπάρχει και κάποια τεντική σφαίρα. Γιατί αυτό επηρεάζει και την οικογένεια κτλ. Εμείς ε, λοιπόν προσπαθούμε βάσει του ορισμού να δούμε κατά πόσο εφαρμόζονται σωστά οι αρχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταία ερώτηση. Η Ανελίζελ Τότσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που δεν ήμουν ε, νωρίτερα εδώ στην αίθουσα. Παρακολουθούσα ωστόσο θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις για τον Ευρωπαϊκό Συντονισμό, όπως και κάποιοι συνάδελφοι. Κάποιοι από εσά είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα FIU σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρχει καλύτερη ε, μια ομάδα, μια υπηρεσία διέξου οικονομικού εγκλήματο, να υπάρχει καλύτερο συντονισμό. Και ακούσαμε και τα θέματα ε, χρηματοδότηση πόρων κτλ. Δεν θέλουμε υπερβολικό όγκο πληροφοριών, αλλά πιστεύετε ότι χρειάζεται ε, ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα για ανταλλαγή πληροφοριών για τις συναλλαγές και για τους ε, κατόχους τέτοιων ε, επιχειρήσεων, εταιρεών. Πιστεύετε ότι είναι αποτελεσματικά τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας και θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και όχι τόσο σε επίπεδο χωρών. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο για να απαντήσει. Ο κύριος Δεκόστερ. Πάρα πολύ σύντομα μια ευρωπαϊκή μονάδα για τη συλλογή χρηματοπιστωτικών πληροφοριών θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή επιλογή άμα θέλουμε να έχουμε μια κοινή ανάλυση. Να έχουμε λοιπόν μια τέτοια μονάδα. Όπως και η Eurojust. Η Eurojust απλώς βάζει ανθρώπους γύρω από ένα τραπέζι, συζητούν και μπορούν να χαράξουν μια στρατηγική. Το ίδιο θα συνέβαινε με μια τέτοια μονάδα χρηματοπιστωτικών πληροφοριών. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάτι σαν την Όλαφ κάτι τόσο μεγάλο όπως η όλοφα, αλλά χρειάζεται να υπάρξει κάποιος τέτοιος φορέας. <clears throat> Ένα παράδειγμα σας δώσω μοναχα τον Ιούνιο, μαζί με τη Γαλλία, αποφασίσαμε και κατανοώντας ότι πρέπει να συνεργαστούμε, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι στα θέματα τρομοκρατίας, αποφασίσαμε να έχουμε μία μονάδα <clears throat> που είναι επάγρυπνη 24 ώρες το 24ωρο και 7 μέρες τη βδομάδα. Η... Δεν έγινε τίποτα. Δεν υπήρξε κάποια απόφαση για συνεργασία με τη Γαλλία. Θέλαμε να κάνουμε κάτι προληπτικά για να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε <clears throat> αίτηση. Τελικά γίνανε όλα στη συνέχεια. Αλλά ήμασταν έτοιμοι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κάτι το οποίο θα αναπτύξουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν ξέρω αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καταφέρει να αλλάξει την οτροπία, αλλά αυτό είναι το βασικό, να αλλάξει την οτροπία του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μοντανιέ, θέλετε να πείτε κάτι για όλα αυτά. Όχι, δεν έχω κάτι να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα έχουμε τα 20 δεύτερα για την ερώτηση της κυρίας Γκόμες. Και το κύριο Ντεκλάης. Είπατε για τα λάθη του καφίνου και για τον Παναμά και γιατί όχι και για την Αγγόλα. Γιατί γίνονται αυτά τα λάθη. Ε, το λάθος γίνεται σαν παράδειγμα στα πλαίσια της τέταρτης οδηγίας για το ξέπλυμα που επιτρέπει εμείς να ψάχνουμε τον διευθυντή της εταιρείας και όχι αυτόν που ωφελείται τελικά από την δημιουργία της εταιρείας. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ο κατάλογος των φορολογικών παραδείσων είναι επίγον αυτό. Και η ομάδα οικονομικής δράσης είχε έτσι και αλλιώς αναφερθεί σε αυτές τις χώρες και μειώνεται ο αριθμός που, των χώρων που ήταν στον κατάλογο. Ένα παράδειγμα, το Μονακό βγήκε από τον κατάλογο. Το άρθρο 1 όμως που επιτρέπει κανείς να μην είναι μόνιμος είναι ότι μπορεί να έχει λογαριασμό αν έχει ένα, ε, ένα λογαριασμό ηλεκτρικού ή λογαριασμό ε, νερού. Για να πετύχει κανείς το Μονακό ακόμα και θύωρος αρκεί. Κώστα, θέλω να προσθέσω κάτι ως ε, απάντηση. Υπάρχει σε αυτόν τον κατάλογο μια χώρα που ψάχνω συνέχεια επιματέω και ίσως το κοινοβούλιο μπορεί να κάνει κάτι. Γιατί η πολιτεία του Delaware στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκεται στον κατάλογο των φορολογικών παραδείσων. Γιατί το Delaware είναι η έδρα της Μοσέκ Φονσέκα, λέει ο κ. Κλές. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα κενά που γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό. Φαντάζομαι ότι και οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να δράσουν στη δική τους χώρα καλύτερα από ότι οι Παναμί, Παναμέζοι εισαγγέλεις. Αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε αν ισχύει. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν στους, στα τέσσερα μέλη του πάνελ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπατε, πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, τις οποίες πρέπει να αξιολογήσουμε. Σα ευχαριστώ για την, τους συναδέλφους για την πάρα πολύ μεγάλη πειθαρχία τους στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης και θέλω να σας προσθέσω ότι την Τετάρτη στις 11 η ώρα θα έχουμε τον καθηγητή Ιωσήφ Στίγλιτς, τον βραβευμένο με Νόμπελ, ο οποίος ήταν και επικεφαλής των εμπειρογνωμόνων της κυβέρνησης του Παναμά για τα Panama Papers. Θα έχουμε περίπου μια μισή ώρα στη διάθεσή μας με τον καθηγητή Στίγλιτς. Και επίσης στις 7 Δεκεμβρίου θα έχουμε τον κύριο Μοσκοβίτσι και την ε, Προεδρία του της Σλοβακίας και της ε, Μάλτας, δηλαδή την προηγούμενη και την επόμενη Προεδρία και το 2017 θα προχωρήσουμε στα επόμενα ερευνητικά βήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνω τη συνεδρία. Σας ευχαριστώ και τους διερμηνείς και σας εύχομαι σε όλους καλό βράδυ. Ένα, ένα λεπτό μόνο καθυστερήσαμε.